Buenas tardes. Good afternoon, everybody. Please be seated. Please be seated. Παρακαλώ, καθίστε, λέει ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Please be seated, dear colleagues. Συνάδελφοι. Ναι, ναι, ναι, ξέρω ότι είχαμε πάρα πολύ δουλειά από τότε που ξεκινήσαμε. Από το χάραμα και ήταν πάρα πολύ έντονο η συζήτησή μας, αλλά παραγωγική, οπότε παρακαλώ προσέξτε και κάντε ησυχία. Intense morning session and then the joint... Είχαμε μια φορτισμένη συνεδρία στο πρωί και κατόπιν είχαμε την κοινή συνεδρία μέχρι τι 2.30 με την ΚΟΝΤ ε, και τώρα αλλάξαμε την αίθουσα και θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ο πύχης είναι ψηλά, οπότε σας παρακαλώ συνεργαστείτε ούτω ώστε να τα πάμε τόσο καλά όσο το πρωί. Έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων. Τώρα με την Eurojust όπου θα έχουμε παρουσίαση του θεματολογίου της υπηρεσίας για αυτή μας την απογευματινή συνάντηση. Όλα αυτά στον τομέα της συνεργασίας για την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η Eurojust και θα μας παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους οι εκπρόσωποι και έχουμε ως ε, προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Eurojust, τον κύριο Λάντισλαβ Χάμαρν. Ως ε, συνήθως θα γίνει ένας πρώτος γύρος ερωταπαντήσεων εκ μέρους των ε, συντονιστών και των ε, προσώπων των πολιτικών ομάδων και κατόπιν οι υπόλοιποι συνάδελφοι αν θέλουν να λάβουν τον λόγο. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε το χρονοδιάγραμμα, τα χρονικά μας πλαίσια, διότι έχουμε δεν έχουμε πάπυρον ε, μπροστά μας για να τη συζητήσουμε ε, την Eurojust, αλλά 45 λεπτά. Γιατί στη συνέχεια έχουμε την περισσή της Λισαβόνας για ε, την παρακολούθηση ναρκωτικών και τοξικομανίας και στη συνέχεια έχουμε την Αστυνομική Ακαδημία, την ΣΥΠΟΛ της Βουδαπέστης. Όλα αυτά με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών που θα μας πούν τι γίνει, οπότε παρακαλώ να τηρήσετε το χρονικό πλαίσιο. Πάμε τώρα. Στον εκπρόσωπο της ε, Eurojust που τον καλωσορίζουμε για να μας ε, παρουσιάσει το τι γίνεται όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της υπηρεσίας τους κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος κλπ. Τι γίνεται δηλαδή σε επίπεδο ε, συνεργασίας για την ποινική δικαιοσύνη. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ στην συνεδρίασή σας και με την ευκαιρία να σας συγχαρώ όλους ε, για την εκλογή σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει να ε, πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια θεωρούμε ότι είστε στρατηγικός εταίρος γιατί μας ε, στηρίζετε, μας βοηθάτε στο έργο μας και σας ευχαριστούμε για όλη σας αυτή την ε, βοήθεια στο παρελθόν. Οπότε βεβαίω και περιμένουμε πώς και πώς την συνεργασία μας τα μέσα επόμενα χρόνια. Ονομάζομαι Λάντισλαβ Χάμπρον. Είμαι ο πρόεδρος ε, της Eurojust και επίσης στη χώρα μου την Σλοβακία είμαι εισαγγελέα. Οπότε έχω αναλάβει να σας παρουσιάσω το έργο του οργανισμού της υπηρεσίας μας για να δούμε τι γίνεται σε διάφορες χώρες από πλευράς πρακτικής και σήμερα σας προσφέρω το έργο της Eurojust. Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες μας. Όπως είπε ο πρόεδρος, θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Πρώτα-πρώτα, Κατα πολέμηση της ε, τρομοκρατίας και το Μητρό για την της ε, τρομοκρατίας, για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ε, διοκτικών και δικαστικών αρχών για την τρομοκρατία. Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή και τέλος θα δούμε τις σχέσεις μας με κάποιες τρίτες χώρες και θα πούμε γιατί αυτό είναι σημαντικό για την δικαστική συνεργασία. 66% από ό,τι γνωρίζω στην Επιτροπή σας είναι τα καινούργια μέλη. Οπότε, να σας πω με απλά λόγια ποια είναι η υπηρεσία μας. Είναι η μόνη υπηρεσία δικαστικής εργασία σε όλο τον κόσμο. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Άρα είμαστε μοναδικοί. Συνεργαζόμαστε με περίπου 100 εισαγγελείς σε 28 κρατούν μέλη και 6 τρίτες χώρες. Όλοι συστεγαζόμαστε και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο ε, με contact points, με σημεία επαφής παντού σε μια ε, κράτη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διασυνορική συνεργασία γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι θα πρέπει να έχουν έγκαιρα αποδεικτικά στοιχεία οι εισαγγελίε, ούτω ώστε να μπορούν να φυλακίσουν τους εγκληματίε. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα ε, από την Αυστρία. Πρόσφατα είχαμε μια υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων. 22 ήταν οι ύποπτοι και 139 όπλα κατεσχέθησαν. Αυτά θα πήγαιναν ε, σε διάφορες μαφίες Οπότε εμείς εξασφαλίσαμε το πώς η παρακολούθηση των τηλεφώνων θα μπορεί να την επικληθεί ο αγγελίας εκεί ε, ως αγνιωπητικό στοιχείο. Είχαν γίνει και τελικά χρησιμοποιήθηκαν στην Ιταλία. Ε, εκεί παραδείγμα στη δοσυνή. Οπότε θα έπρεπε να κάνουμε και την μεταφορά ε, από τη μία χώρα στην άλλη. Πέρσι επίσης είχαμε την εκτέλεση πάνω από 700 ενταλμάτων σύλληψης, τα οποία αποτελούν την ε, νομική βάση για σύλληψη κάποιου που μένει κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, θα μπορούσε κανείς να πει γιατί έχουμε τόσα πολλά που πρέπει να εκτελέσουμε. Μα ε, αυτά ζητήθηκαν από δικαστές και εισαγγελίες γιατί πολλές φορές ζητούνται στοιχεία, επιπλέον στοιχεία, ένα σωρό στοιχεία για το εν λόγω έγκλημα, για τις συνθήκες κράτησης, τις φυλακές και όλα αυτά γιατί αυτά τα στοιχεία πολλές φορές λείπουν από τα ευρωπαϊκά εντάλματα. Οπότε θεωρείται ως πρακτική λύση εμείς να δώσουμε αυτές τις ε, πληροφορίες όσον αφορά την χώρα τις οποίε οι ιδιωτικέ αρχές επιλαμβάνονται και το κάνουμε γρήγορα. Τώρα από πλευράς επιμελητίας, από πλευρά ε, των ομάδων μας ε, βοηθήσαν πάνω από 200 ε, ομάδες που διεξέγουν δικαστικές έρευνες όπως και στο Μπολίνο που είχαμε συνεργασία τριών χωρών και εκεί έγινε συντονισμός ε, πάρα πολύ σημαντικός για την Ευρώπη της Ντράγκετα και τελικά είχαμε 84 συλλήψεις σε όλο τον κόσμο και κατάσχεση ε, τεσσάρων τόνων κοκαίνης αλλά και αντικειμένων αξίας 2 εκατομμυρίων οπότε α, ένα δις κόστιζε αυτή η κοκαίνη που κατεσχέθη τόσο κοστίζει στην ε, αγορά Κανεί θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί θα πρέπει να επενδύονται χρήματα σε αυτές τις κοινέ δικαστικέ έρευνε, μα διότι ο κόσμο, αν ε, πρέπει και αν χρειάζεται τη συνεργασία, πρέπει να ανταλλάξει πληροφορίε, να γίνουν ταξίδια, ε, όλα αυτά κοστίζουν. Επίση, χρειάζονται και μέσα τεχνική υποστήριξη για την ασφάλεια των επικοινωνιών. Στην περίπτωση, στην υπόθεση που σα είπα, εμεί χρηματοδοτήσαμε αυτέ τι κοινέ ομάδε. Ε, ύψους 180.000 ευρώ. Και βλέπετε όμως τι αποτέλεσματα αποσπάσαμε εις όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Να ένα παράδειγμα του πόσο αποδίδουν οι επενδύσεις. Επίσης, για κατασχέσεις και για ε, συλλήψεις όταν γίνονται ταυτόχρονα από τα κράτη-μέλη και χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία, το κάνουμε αυτό και είχαμε κάποια υπόθεση τον Ιούλιο φέτος όπου είχαμε 28 έρευνες σε εταιρείε, σε οικίες, σε Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, ε, Βοσνία, Ριζεγοβίνη και αλλού και σε αυτή την περίπτωση ε, βοηθήσαμε για μια υπόθεση ξεπλήματος χρήματος. Όλα αυτά τα συντονίσαμε από την Χάγια, από την έδρα μας. Σε πραγματικό χρόνο βοηθήσαμε τους επιτόπου συναδέλφους ε, για συλλογή στοιχείων κλπ. Και έτσι οι σχετικές χώρες μπόρεσαν να προβούν σε κατασχέσεις ε, πάρα πολλών ακριβών ε, αντικειμένων όπως ακόμα και πολιτών αυτοκινήτων εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης ένα πληρωμένο δολοφόνο από τη Σερβία, βοήθησαμε να τον συλλάβουν. Είχε κάνει σε Άμστερνταμ, Βελιγράδι, Βουδαπέστη ε, δολοφονία και συνελήφθη στην Τσεχία. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να βοηθήσουμε να υπάρχει επικάλυψη στα διαφορετικά αντάλληλα, γιατί όλες οι χώρες θέλανε να τον συλλάβουν και να τον πάνε στην δικαιοσύνη. Αλλά εμείς ε, κρίναμε το ποια είναι η καλύτερη χώρα, ο καλύτερος τόπος να συλληφθεί, πού υπάρχουν τα πιο γερά αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε αναλύσαμε όλες τις πληροφορίε που είχαμε, όλα τα πραγματικά περιστατικά από όλε τι χώρε και έτσι τελικά ε, τον στείλαμε στην Ουγγαρία για να παρενθέσει τη δικαιοσύνη. Θα μπορούσα να συνεχίσω με ένα σωρό παραδείγματα, αλλά πιέζει ο χρόνος. Πάντως με δύο λόγια, αυτό που κάνουμε είναι το ότι βοηθούμε τους εισαγγελείς. Σε ενωσιακό επίπεδο βοηθούμε τους συναδέλφους επομένως σε όλες τις χώρες. Και θέλουμε να δίνονται πρακτικές λύσεις για τα πρακτικά χειροπιαστά προβλήματα. Έχουμε ένα σωρό στοιχεία που δείχνουν το πόσο έχουμε πετύχει οπότε και εσείς μπορείτε να δείτε τώρα σε αυτή την διαφάνεια ότι κάθε χρόνο διεκπεριώνουμε και περισσότερες υποθέσεις. Δεν επιβάλλουμε τίποτα στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για συνεργασία που γίνεται μόνο αν θέλουν να μας παραπέμψουν μια υπόθεση και όταν έχουν κάποια δύσκολη υπόθεση αποφασίζουν ότι ναι, θα πάμε και θα απευθυνθούμε για βοήθεια στην Eurojust. Έτσι έχουμε προχωρήσει, 22% νέες υποθέσεις το 18%. Και δυστυχώς η προκοδότηση δεν αντιστοιχεί στην αύξηση των υποθέσεων, κάτι το οποίο μας αποκτεύει πάρα πολύ. Είναι αντικίνητρο για τους εισαγγελείς που βοηθάνε. Αλλά χωρίς χρήμα δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Οπότε, εμεί ε, θέλουμε όπω και πώ να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κρατη αλλά θέλουμε να μα βοηθήσετε όχι για να ε, αποθεωθεί η υπηρεσία μα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε του αδέλφου που εργάζονται κατά του ιδιωτικού εγκλήματο στη χώρα του. Να ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς βοηθούμε Βεβαίω προσπαθούμε να γίνουμε στο λένε και καλύτεροι και προσπαθούμε να δέχτουμε από τα λάθη μα. Να, ένα τομέα που θέλουμε να βελτιωθούμε είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών όσον αφορά τι υποθέσει τρομοκρατία ή καταπολέμηση τρομοκρατία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το μητρό για την εντόπιση της τρομοκρατίας. Ξεκίνησε την πρώτη Σεπτεμβρίου, πριν από λίγε μέρε. Γιατί χρειάζεται, τι είναι αυτό ακριβώ, διότι οι τρομοκράτε ω εγκληματίε κινούνται όλο και περισσότερο από μια χώρα στην άλλη. Και ω αποτέλεσμα υπάρχουν όλα και περισσότερε πιθανότητες ότι η ίδια συμμορία ή ο ίδιος τρομοκράτης ε, υπόκειται έρευνα σε πάνω από μία χώρα. Οπότε για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός αυτών των ερευνητικών προσπαθειών και έχουμε πέντε παραδείγματα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέεται μία έρευνα με την άλλη. Διότι εάν κανείς κάνει την διασύνδεση και συνδυασμό των ερευνών, αποφασίζει κανείς αν χρειάζεται να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση και επίσης ε, χρειάζεται να διεξαχθεί από κοινού ή εν λόγω κάθε φορά έρευνα και αυτό το μητρό ε, μπορεί να μας ε, βοηθήσει να δούμε το ότι κάποιος τρομοκράτης ανήκει σε μια συμμορία τρομοκρατική ομάδα που δράσει άλλη χώρα και ε, έτσι μπορούμε να σπάσουμε τη δικτύωσή τους και μπορούμε να επιβάλλουμε ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις. Μπορεί τα αποτικά στοιχεία που συνελέξαν σε μια χώρα μπορεί να ωφελούν άλλη χώρα στην προσπάθειά της που κάνει την έρευνα για τον ίδιο ύποπτο. Οπότε αυτό το αρχείο, αυτό το μητρό ε, αποτελεί εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και υλικών πόρων και ε, να μην έχουμε επικάλυψη. Έτσι, οι κατασχέσεις και οι συλλήψεις μιας χώρας δεν θα αποτελούν φραγμό σε ποινική δίωξη ή σε έρευνα άλλης χώρας. Και τελευταίο, αλλά σημαντικό, σύμφωνα με το άρθρο 50 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης ουδής μπορεί να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ή να καταδικαστεί δύο φορές για το ίδιο έγκλημα. Οπότε με τη διασύνδεση των υποθέσεων έτσι προστατεύουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε, συνεχίσουμε τα κρατημέλη, φτιάξαμε αυτό το μήτρο, αυτό το αρχείο και έτσι τα κρατημέλη μας ε, κοινοποιούν τις πληροφορίες, οπότε τώρα έχουμε ένα εργαλείο για μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Οπότε, τελευταίο αλλά σημαντικό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων ε, είναι τώρα σε υψηλά ε, στάνταρ μέσω αυτού του ποινικού μητρώου. Για να δούμε τώρα, έχουμε ένα σωρό προκλήσεις για το μέλλον ως υπηρεσία και ως ε, δικαστές και εισαγγελείς όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, όλου του κόσμου. Το θέμα είναι η ψηφιοποίηση και το άλλο είναι η παγκοσμιοποίηση. Οπότε για την ε, ψηφιακή τεχνολογία πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι όλα είναι και περισσότερες πληροφορίες μας έρχονται και πολλά και περισσότερες υποθέσεις. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι αυτές έρχονται με διαφορετικά πρωτόκολλα, διαφορά στο περιεχόμενο, κάθε χώρα έχει το δικό της στυλ, οπότε μετά την ε, λήψη των ε, δεδομένων Συνήθω χρειαζόμαστε βοήθεια για να τα επεξεργαστούμε, μεταφράσει. Αυτό τρώει, πάρα πολύ χρόνο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε διασταύρωση των πληροφοριών. Μόνο έτσι. Αλλά όλα αυτά πολλέ φορέ γίνονται με μη αυτοματοποιημένου ε, τρόπου. Για να μπορούμε τέλο πάντων να αποσπάσουμε κάποια συγκεκριμένα ε, απτά αποτελέσματα και να αξιοποιηθούν οι βάσει δεδομένων. Οπότε, γι' αυτό και εμεί προτείναμε ως λύση έναν νέο τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων με συνεργασία της Eurojust με τα κράτη-μέλη. Όμως είναι σημαντικό αυτή η ανταλλαγή στοιχείων ε, να γίνεται και με τη Europol, τη Frontex, ε, την καινούργια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν είναι δυνατόν ο καθένας να δρά από το πύργο του. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε για να συνδυάζουμε τις προσπάθειες. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό διεθνές έγκλημα. Έτσι θα κάνουμε τη διαφορά. Το με αυτά στου υπουργού δικαιοσύνη, τι προτάσει ε, μα. Είπαν ότι μα υποστηρίζουν ε, οπωσδήποτε. Και να, έχει γίνει επομένω ένα ουσιαστικό βήμα προ την επιθυμητή κατεύθυνση. Και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και η συνεργασία μας με τις διοικητικές αρχές ε, που φυσικά έχουν προχωρήσει, έχουν κωδικοποίηση για την ανταλλαγή των πληροφοριών και θα πρέπει ότι κάνουν διοικητικέ αρχές να τα κάνουμε και εμείς στον τομέα της δικαιοσύνης. Δεν είναι λογικό να προστατεύεται ένα αγαθό, ένα δικαίωμα, κάτι σε αστυνομικό επίπεδο, αλλά εμείς να μην κάνουμε στο δικό μας επίπεδο το ίδιο σε επίπεδο δικαιοσύνη Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι δύο του ίδιου νομίσματος γίνεται η σύλληψη από την διοικητική αρχή και εμείς ασκούμε την ε, δίωξη ούτω ώστε να φυλακιστεί ο ένοχος. Ε, βέβαια, χρειάζονται κάτι παραπάνω από στοιχεία, από πληροφορίε. Χρειάζονται κάποιες, ε, κάποια, κάποια βάση από δικά στοιχεία. Τέλο πάντων, ε, όλα αυτά τα συζητούμε και θα τα συζητήσουμε στι 10 Δεκάτου στο Συμβούλιο των Βρυξελών. Με το θέμα τη ποινική δικαιοσύνη τον ψηφιακό κόσμο, στη διαρχή εποχή, ε, και σε αυτή την συνάντηση είστε όλοι προσκεκλημένοι. Τώρα, άλλο θέμα, άλλο μέτωπο είναι η παγκοσμιοποίηση. Οπότε διαπιστώνεται ότι κινούνται όλο ένα και περισσότερο διεθνώ οι ε, ύποπτοι, οπότε χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερα στοιχεία, όλο ένα και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία από τρίτε χώρε. Ε, για αυτό, ότι και κάποια χρόνια έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο ε, με επαφές μας στις τρίτες χώρες και ε, έτσι καλύψαμε 1.300 υποθέσεις που αφορούσαν τέτοιες ε, τρίτες χώρες. Οπότε έχουμε αύξηση 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και τώρα έχουμε 11 συμφωνίες ε, συνεργασίας και έχουμε επαφές με 49 χώρες. Και έχουμε τη διαφορά ότι σε όποια χώρα δεν, δεν ισχύει κάποια συμφωνία έχουμε αυτά τα σημεία επαφής ε, για να κάνουμε μια συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών. Όχι τόσο συστηματικά όσο με τις ε, διεθνείς συμφωνίες. Οπότε, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να παγιωθούν ε, οι σχέσεις μας με αυτές τις χώρες Δυτικά Βαλκάνια, Λατινική δηλαδή Αμερική και όχι μόνο. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα αυτή η πολιτική και αυτά θα τα πούμε στη σημερινή μας συνέντευξη όταν ήρθε να συζητήσουμε για τις σχέσεις με την ε, Σερβία όταν θα, έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την σχετική συμφωνία όπου βέβαια θα χρειαστεί και η δική σας συνεργασία. Α, Βλέπω ότι ξέχασα να παρουσιάσω κάποιες διαφάνειες και συμπαθάτε με. Εδώ, αυτή η διαφάνεια απλώς... Α, αυτό αποδεικνύει ότι δεν μπορεί κανείς να τα κάνει όλα ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, τώρα μπορώ να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσίασή μου και ελπίζω ότι η σημερινή συνάντηση είναι η αρχή μιας μεγάλης διαδρομής και με τις προσπαθειές μας θα υλοποιήσουμε την συνεργασία με τις τριτές χώρες και ότι θα ξανασυζητήσουμε το τι γίνεται με την ποινική δικαιοσύνη ε, και την ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει να σας πω ότι ξέρουμε ότι χρηματοδοτούμεθα από τον δημόσιο κορβανά και ότι είμαστε υπόλογοι σε εσά. Πάντως το σημαντικό είναι ότι έχουμε το ίδιο καθήκον να εξυπηρετήσουμε και να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους που και εσείς αυτό θέλετε να πετύχετε, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη στην ε, Ευρώπη. Ευχαριστούμε για αυτή την εξαιρετική ε, παρουσίαση και για το τηρήσατε το χρόνο. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε τους συντονιστές και μετά υπάρχουν και κάποια μέλη της Επιτροπής μας που έχουν ζητήσει το λόγο. Σας έχουμε σημειώσει. Όμως, δεν βλέπω το συντονιστή του ΕΛΚ, οπότε θα πάρω εγώ πρώτος τον λόγο εκ μέρου. Ε, μάλλον θα περάσω εγώ ε, και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σίπελ, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ε, κάνω κάποιε παρατηρήσει και δύο ερωτήσει. Η παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι έχω πιστεί ότι δεν είναι κανεί αποτελεσματικό στην, στον τομέα τη ποινική δικαιοσύνη χρειάζονται και αστυνομία και δικαιοσύνη να λειτουργούν σωστά και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του. Οπότε εδώ υπάρχει σίγουρα περιθώριο βελτίωση και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρατήρηση, απλή. Μετά, έχω δύο ερωτήσει. Θυμάμαι τις τελευταίες, τα τελευταία δέκα χρόνια σε διάφορου τομεί είχαμε συζητήσει για τι συνθήκε που επικρατούν στι φυλακέ. Κατά τη γνώμη σα, Συμφωνείτε με την άποψη ότι χρειάζονται αλλαγές και ενδεχομένως κάποια βήματα εναρμόνισης. Και έχω και ένα δεύτερο ερώτημα για το αντιτρομοκρατικό μητρό. Βλέπω πόσο ένα τέτοιο μητρό θα μπορούσε να βοηθήσει και γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο μητρό. Έχουμε όμως προβλήματα πολύ συχνά με τους ορισμούς. Και όσον αφορά τον ορισμό του τρομοκράτη, του ποιος είναι τρομοκράτης. Έχετε καταφέρει εσείς να καταλήξετε σε ενιαίο κοινό ορισμό και για τα 28 κράτη-μέλη ή μήπως έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς ορισμούς. Οπότε ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το κατάλογο, σε αυτό το μητρό που θεωρούνται τρομοκράτες σε μία χώρα ενώ σε άλλη χώρα όχι. Και τι σημαίνει αυτό για την αντιτρομοκρατική δουλειά. Ευχαριστώ. Η Σόφη Ιντβελτ εκ μέρους της ομάδας Renew αν θέλετε το λόγο. Ξέρω ότι και ο συνάδελφος ο κύριος Χουκ θέλει να πάρει το λόγο, αλλά έχετε εσείς πρώτοι το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα και θα δώσω το λόγο και μετά στους συναδέλφους. Ε, δύο ερωτήσεις έχω να θέσω. Ε, άργησα λίγο να έρθω, ίσως να το αναφέρατε, αλλά δεν το άκουσα. Πρώτον, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το ρόλο της Eurojust στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς έχετε κάνει, ποια είναι εν γέννη η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ερώτημα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου η δικαστική εξουσία δεν ανταποκρίνεται αν θέλετε, ε, στα πρότυπα ποιότητα που ε, οφείλει να τηρεί κάθε κράτος μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, η Πολωνία. Ε, το, μάλιστα η πολωνική δικαιοσύνη έχει ανασταλεί η ιδιότητά της, η συμμετοχή της στο δίκτυο δικαστικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόβλημα, πώς, είναι η συνεργασία σας με τέτοιε χώρε. Ευχαριστώ. Βλέπω η πράσινη, η κυρία Τρίκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να θέσω και εγώ αυτό το ζήτημα που έθεσε η κυρία Ιντβελτ, το ζήτημα της αμοιβαία εμπιστοσύνης, που είναι σημαντικότατη για την συνεργασία αυτή. Έχουμε φυσικά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Πολωνία. Έχουμε και την σύγκρουση μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας λόγω της γερμανικής απόφασης να μην ε, ε, συνεργαστεί ε, όσον αφορά την ε, παράδοση των Καταλανών αποσχιστών. Πώς επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα τη δική σας δουλειά και θα μπορούσατε να μας δώσετε ίσως κάποια παραδείγματα όπου κάποια κράτη-μέλη ε, μπορούν ε, ε, που έχουν μάλλον υψηλά διαδικαστικά εχέγγυα, πώς γίνεται να, να, να χειρίζονται υποθέσεις με χαμηλότερα πρότυπα. Και μετά υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά τον προϋπολογισμό. Υπάρχει απειλή από τη μείωση. Ποιος, θα είναι ο αντίκτυπος των μειώσεων στον προπολογισμό σα και για τι τρίτε χώρε και τη συνεργασία μαζί του. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα, τα προσωπικά δεδομένα, αφού φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουν να, υπο, να υπόκειται σε ένα καθεστώ προστασία όπω αυτό που ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω συντονιστέ από το ID και το ECR. Φαντάζομαι όμω ότι εσεί, συνάδελφε, του εκπροσωπείτε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ ε, και για την παρουσίαση και για την ε, στατιστική που μας διαβάσατε, τα στατιστικά στοιχεία που μας δώσατε για πέρσι. Πρώτο, βεβαίως η Eurojust θα πρέπει να είναι καλός εταίρος για τα κράτη-μέλη, γιατί αν, εφόσον υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι, τότε προφανώς υπάρχει και μια αρνητική όψη αυτού του νομίσματος, όπως για παράδειγμα το να μεταφέρονται τόνοι κοκαίνης από τη μία χώρα στην άλλη. Οπότε είναι προφανές ότι χρειάζεται καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της Eurojust. Βλέπω ε, από τα στατιστικά στοιχεία ότι από το 2014 στο 2018 υπάρχει ε, αύξηση ε, των, των, συλλήψεων και των υποθέσεων που αφορούν την τρομοκρατία. Και φέτος. Ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία και την μαζική μεταναστευτική κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 5-6 χρόνια στην ε, Ευρώπη. Πώς συνδέονται η τρομοκρατία και η μετανάστευση. Επίσης, άμα δούμε τα στοιχεία από τα διάφορα κράτη-μέλη, όπως ε, κάποιος συνάδελφος ε, αναφέρθηκε στην Πολωνία, ε, άμα, δούμε, άμα κοιτάξουμε βεβαίω και την Σουηδία, υπάρχει, υπάρχει μεγάλη διαφορά στους αριθμούς τρομοκρατικών επιθέσεων. Και άμα, επιθέσεων. Και άμα δει κανείς και τις μεταναστευτικές ροές, το πού πηγαίνουν δηλαδή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ε, τότε επειδή εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας όπως είστε εσείς, ίσως θα μπορούσατε εσείς να μας δώσετε κάποια περισσότερα στατιστικά στοιχεία και να μας πείτε ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο φαινομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάντισον. Okay. Ε, Εσείς κύριε συνάδελφε από την Ιταλία, συγγνώμη που δεν σας δίνω το λόγο. Καλησπέρα συνάδελφε και εσάς ε, ευχαριστούμε κύριε για την ε, παρουσίαση. Σύντομη ερώτηση των Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η πρώτη συνάντηση συντονισμού Eurojust με χώρες Δυτικής Αφρικής. Κατόπιν κάποιων τρομοκρατικών ενεργειών. Ερωτώ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν συνθήκες για μια συνεργασία ούτως υπήν συστηματική, πάγια, μόνιμη για αυτά τα θέματα με εκείνε τι χώρε. Με για κάποια θετική συνεργασία ακριβώς με αυτές τις συμφωνίες που ήδη έχετε συνάψει με κάποιες τρίτες χώρε. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Κύριε ευχαριστώ. Δεν έχω ε, καταλάβει ακριβώς ε, τι συμβαίνει με το αντιτρομοκρατικό μέτρο ε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερε πληροφορίες. Πώς μπορεί κανείς να ενταχθεί αυτή. Υπάρχει κάποια βάση δεδομένων. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν διωχθεί ή είναι απλώ ύποπτοι για συμμετοχή στη δημοκρατία. Τι είδους πληροφορίες επίση ανταλλάσσονται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Και αν ναι, ποια είναι η νομική βάση για να γίνεται κάτι τέτοιο. Μήπω ε, θα ε, μπορούν ε, τα στοιχεία αυτά να διορθώνονται ή και να αφαιρούνται στη συνέχεια. Για την πρωτοβουλία Digital Criminal Justice. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το Project Sirius που ε, χρηματοδοτείται από την Κομισιόν για την εξωτερική πολιτική. Ε, λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση που λαμβάνουν ε, οι επαγγελματίες του χώρου για την νομική συνδρομή, γιατί χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένα νέο project. Υπήρχαν κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονταν από τα υπάρχονταν. Και τέλος, για την συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Μπορείτε να μας περιγράψετε το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε εσά και τη Λιβύα και ανάμεσα σε εσά και το, και, και το Αφγανιστάν και ποια είναι, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτές της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Για τους συντονιστέ των πολιτικών ομάδων ολοκληρώσαμε και αν μου επιτρέπετε εκεί. Ε, δεδομένου ότι το χρονικό πλαίσιο είναι ακόμα πιο σφιχτό από σήμερα το πρωί, θα ήθελα να δώσουμε ένα λεπτό ακόμα σε πέντε ακόμα μέλη που θα θέλουν να πάρουν το λόγο και μετά θα μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση με τις απαντήσεις σας, ακόμα και αν ξεπεράσουμε το χρονικό ε, διάστημα που προβλέπετε. Ο κύριος Κέρνερ έχει τώρα από τη Ρενιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την σημαντική δουλειά που κάνετε. Δύο ερωτήματα έχω να απευθυνώ. Τα αγγίξατε τα θέματα αυτά, αλλά και εμένα μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η μείωση στη χρηματοδότηση στο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς αυτή η μείωση θα επηρεάσει αρνητικά τη δουλειά σας και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την ε, λειτουργία του EPPO, πώ θα επηρεάσει το Eurojust. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία και πολύ σύντομο. Σε ευχαριστώ πολύ από την Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, η επόμενη μελετητρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάναν. Έχω δύο γρήγορες ερωτήσεις να κάνω για την τρομοκρατία. Καταρχάς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την ε, κατάσταση την τρομοκρατία, η τρομοκρατία στα κράτη-μέλη ξεκαλουθεί να αυξάνεται διπλή για δεύτερη συνεχή χρονιά οι απειλέ. και τα κράτη-μέλη παίρνουν στα σοβαρά τα, τις απειλές αυτές χρησιμοποιούν πιστεύετε όμω τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και τι άλλα μέτρα μπορούν να λεφθούν σε επίπεδο άμα Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά του Ευρωπαίου πολιτε που έχουν διαπράξει εγκλήματα σε σχέση με την ISIS. Από ό,τι μας είπατε, δημιουργήθηκε σχετική απόφαση μάλλον την, ε, το Σεπτέμβριο και το εργαλείο, συγγνώμη. Ε, ποιο, ποιο μπορεί να είναι ο αντίκτυπο του εργαλείου αυτού σε ό,τι αφορά το συντονισμό των δράσεων μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αν γίνει το Brexit, πώς θα επηρεάσει αυτό τη Eurojust, τι θα γίνει με τις πολλαπλές ε, περιπτώσεις και υποθέσεις της ε, Βρετανίας ή πολλές ε, υποθέσεις στα άλλα κρατημέλη που σχετίζονται με τη Βρετανία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρίκμο. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δύο πράγματα θα ήθελα να ξέρω. Τι είδους συνεργασία Ε, υπάρχει για τους ε, μαχητές του ISIS που έχουν επιστρέψει και τι είδους συνεργασία υπάρχει από πλευράς ε, των θυμάτων, θυμάτων οργανωμένου κλίματος, τρομοκρατίας. Αναμένουμε την έκθεση εφαρμογής για την οδηγία για την προστασία των θυμάτων και θα ήθελα την δική σας εκτίμηση για την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Η κυρία Κέλλερ. Υποστηρίζω την ερώτηση της κυρίας Πεδίκμαν σε ό,τι αφορά τους ε, αλλοδαπούς μαχητές. Παρακολουθείτε τα άτομα τα οποία έχουν φύγει από την Ευρώπη με ευρωπαϊκή υπηκότητα και σε κάποιες περιπτώσεις και τις οικογένειες τους που ε, διατηρούν συνδέσμους μαζί τους. Και κατά δεύτερον, η ίδια ερώτηση του κ. Κέρνερ σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του προπολογισμού. Πείτε μας, Ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία θα ανακύψουν εάν δεν πάρετε τη χρηματοδότηση την οποία θέλετε. Είδατε ζητάει άλλος ένα το λόγο. Αν είστε σύντομοι όμως. Θα είμαι, θα είμαι σύντομος. Ναι, ναι, ναι δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. και μετά θα μας απαντήσει ο πρόεδρος της ε, Eurojust. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα αριθμητικά στοιχεία για την αύξηση των ε, περιστατικών τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος έχετε επαρκείς ε, πόρους για να αντιμετωπίσετε την αύξηση αυτή και κατά δεύτερον υπάρχει διαφορά μεταξύ κρατών μελών στη συμμετοχή στις δραστηριότητε της Eurojust, γιατί στον πίνακα που δημοσιεύθηκε δεν βλέπουμε διακοπές, διαφορές, συγγνώμη, ε, με κάποια κρατημέλη τα μεγάλα ενδεχομένω να έχουν κάποιες υπόλοιπε αλλά γενικά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα μιλήσω την ε, εθνική μου γλώσσα για να σεβαστούμε και την ε, διαφοροποίηση στην Ευρώπη. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει έλεγχο συνόρων, ε, υπάρχει όμως ε, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής και έχω υπόψη μου τη νομοθεσία της Ιταλίας, της Ουγγαρίας σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ που διευκολύνουν το, τη διακίνηση ανθρώπων στην Ευρώπη. Αν λοιπόν γίνεται σεβαστή μία νομοθεσία σε μια χώρα και σε άλλες όχι. Εσείς εμπλέκεστε, συμμετέχετε και κατά δεύτερον, όταν υπάρχει τέτοιε εγκληματικές δραστηριότητε, εσείς συλλέγετε πληροφορίες για τα οικονομικά δίκτυα που υποστηρίζουν αυτές τις ΜΚΟ. Και τώρα έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ξέρω ότι έχουμε υπερβεί το χρονικό όριο και δεν έχουμε επαρκή χρόνο. Ο επόμενος ε, ομιλητής είναι ήδη στην αίθουσα επικεφαλής ε, της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της ε, ναρκωτικών. Αλλά σας παρακαλώ να απαντήσετε γρήγορα. Yes, uh, many thanks to... Ναι. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις και για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Θα προσπαθήσω ε, να απαντήσω κατά θεματική κατηγορία. Υπήρξε λοιπόν ένα ερώτημα που αφορούσε την αμοιβή εμπιστοσύνη και αν υπάρχει διάβρωση αυτής της εμπιστοσύνης. Και αυτό συνδέεται και με το ερώτημα της κυρίας Ζίπελ που αφορούσε τις ε, συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Πράγματι, βλέπουμε μια μεταστροφή από την αρχή της αμοιβαία ε, εμπιστοσύνης, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα νομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται σε αυτήν ακριβώς την αρχή, την αρχή της αμοιβαία εμπιστοσύνης. Ιδίω λοιπόν μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου φαίνεται να υπάρχει μια ελαφρά μεταστροφή. Εγώ δεν θα το αποκαλούσα διάβρωση της ε, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ε, θα έλεγα όμως ότι ε, πρόκειται για μια αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης. Υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη, αλλά δεν είναι πλέον τυφλή μεταξύ των κρατών μελών και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, τα, οι εκτελεστικές αρχές ε, των κρατών μελών ζητούν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για παράδειγμα τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Από εκεί ξεκινήσαμε για το πόσα τετραγωνικά μέτρα για παράδειγμα θα έχει ένας κρατούμενος στην εκάστοτε χώρα, στην τάδε χώρα. Ε, μιλούσαμε, ε, συνεχίσαμε ε, για τις συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, για την διατροφή των κρατουμένων, μέχρι που καταλήξαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση για το πόσο δημοκρατική, αν θέλετε, είναι η διαχείριση ή κατά πόσο συμβαδίζουν με τις αρχές του κράτους δικαίου τα δικαιϊκά συστήματα των κρατών μελών. Ε, πρόκειται για υποχρεώσεις ε, των ε, κρατών μελών να επαληθεύουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, όλα αυτά τα στοιχεία και εξ αυτού προκύπτει και αυτός, αυτή η αύξηση των ερωτημάτων που θέτουν το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και αυτά τα ερωτήματα πολύ συχνά καταλήγουν στη Eurojust ακριβώς γιατί η Eurojust θεωρείται ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να παράσχει, να παρέχει γενικά τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα στις γλώσσες ε, των κρατών μελών, στη γλώσσα του κάθε κράτους μέλους και με τον τρόπο που ε, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε πολύ εντατική επικοινωνία με ε, διάφορες χώρες. Πρόεδρε, θέλατε να με διακόψετε να μου πείτε κάτι. Όχι, λέει ο πρόεδρο. Απλώ με ενδιαφέρει πολύ το θέμα και σα παρακολουθώ ε, με μεγάλη προσοχή. Μετά, το ερώτημα τη κυρία Ζίπελ αφορούσε τον ορισμό τη τρομοκρατία. Νομίζω ότι για τα κράτη-μέλη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό είναι λιμένο. Τα κράτη-μέλη πλέον έχουν κοινό ορισμό για την τρομοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, δεν υπάρχει συμφωνία για το τι ακριβώς είναι η τρομοκρατία, τι συνιστά ε, τρομοκρατία, τι σημαίνει ο όρος τρομοκρατική οργάνωση. Και αυτός ο ορισμός ε, πράγματι δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Για το ερώτημα που αφορούσε την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, και συγκεκριμένα την κατάσταση στην Πολωνία. Εγώ είπαμε, ε, σας είπα είμαι, είμαι εισαγγελέα. πολιτικός δεν είμαι. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι από την Πολωνία κάνουν ό,τι μπορούν για να μας παρέχουν τη βοήθεια, τη συνδρομή που χρειάζονται ή που ζητούν άλλα κράτη-μέλη. Εμείς δεν έχουμε γίνει μάρτυρες προβλημάτων, ζητημάτων, εμποδίων. Τα πράγματα πηγαίνουν ε, πολύ καλά. Ωστόσο, όπως είπα, λόγω του ζητήματος της εμπιστοσύνης, αυτό πράγματι έχει επιπτώσεις όσον αφορά τις απαιτήσει. Και βεβαίως η έκθεση της Κομισιόν που επέκρινε ε, ορισμένες χώρες ε, χρησιμοποιήθηκε από, ως συγκριτικός δείκτης αν θέλετε για, ε, από ορισμένες εκτελεστικές αρχές όσον αφορά τις ε, παραδόσεις στην Πολωνία. Ε, ε, το, υποβλήθηκαν πολύ περισσότερα ερωτήματα που σημαίνει ότι η πολυνομία αναγκάστηκε να δώσει πολύ περισσότερες απαντήσεις από ό,τι στο παρελθόν σχετικά με την ανεξαρτησία του συστήματος ε, δικαιοσύνης τους. Περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο πραγματικός αντίκτυπος αυτόν που είδατε στην οθόνη για τα επόμενα 7 χρόνια οι περικοπές αυτές είναι μια πραγματικότητα, αν γίνουν πραγματικότητα μάλλον, ε, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα ως Eurojust. Θα πρέπει να ε, βρούμε ε, πόρους, διότι έχουμε λογαριασμούς να πληρώσουμε, ενίκεια, ε, ε, ρεύμα και αυτό που ε, ε, Δυστυχώ θα σημάνει η περικοπή του προπολογισμού μα θα είναι ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την επιχειρησιακή υποστήριξη που το κάναμε, ε, όπως το κάναμε μέχρι τώρα. Δεν θα μπορούμε να παρέχουμε μετάφραση, διερμηνία για εισαγγελεί που έρχονται στην Eurojust για να συζητήσουμε διάφορες υποθέσεις. Πολύ απλά οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρότατες από την περικοπή αυτή του προϋπολογισμού και πεποίθησή μου είναι ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών ε, θα μειωθεί σημαντικά γιατί ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, και στις πολλές, σε πολλά κράτη-μέλη η δικαιοσύνη υποχρηματοδοτείται επομένως δεν θα υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι για να οργανωθεί αυτή η αναγκαία κατά τα άλλα συνεργασία. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιε περικοπέ σε κάποιου τομεί, όμω θεωρούμε ότι δεν είναι ε, η σωστή στιγμή ούτε ο σωστό τομέα για να γίνουν αυτέ οι περικοπέ. Συνεργασία με τρίτε χώρε, προστασία προσωπικών δεδομένων. Εμεί έχουμε συνάψει συμφωνίε συνεργασία με τρίτες χώρες μόνο εφόσον ε, λάβουμε ε, το τελικό πράσινο φως από ε, τους ειδικού επί, επί του ζητήματο της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και αυτό είναι πάντοτε μια από τις βασικότερες απαιτήσει για να συνάψουμε συμφωνία συνεργασίας με τρίτη χώρα. Εμείς πάντοτε ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν το τι ακριβώς θα γίνει με τα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών όταν αυτά μεταφέρονται σε τρίτη χώρα. Και μόνο εφόσον υπάρχουν ε, σωστά και επαρκή εχέγγυα ότι στη χώρα την τρίτη τηρούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μόνο τότε ε, συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες. Γι' αυτό και έχουμε λίγες ε, στον αριθμό τέτοιες. Θα θέλαμε να ήταν περισσότερες, αλλά πάντοτε έχουν απόλυτη προτεραιότητα τα, τα πρότυπά μα όσον αφορά την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Μετανάστευση και τρομοκρατία και διασύνδεση αυτών των δύο. Εμείς στην ε, Eurojust δεν ε, είμαστε οι πλέον αρμόδιοι για να σας πούμε για κάποιες συγκεκριμένες τάσεις, γιατί δεν συλλέγουμε όλα τα δεδομένα από όλες τα κράτη-μέλη. Όλες οι υποθέσεις που παραπέμπτονται στη Eurojust είναι τυχαία αιτήματα όπου υπάρχει ανάγκη να δοθεί βοήθεια σε εισαγγελικές αρχές, δικαστικές αρχές ε, για, τις, ε, ε, για τη μετανάστευση δεν μπορώ να σας πω. Μιλάμε πάντοτε για υποθέσεις όπου έχει κάποιο κράτος μέλος αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και ζητά την υποστήριξη της Eurojust. Εμείς τέτοιες υποθέσεις χειριζόμαστε, ποτέ δεν αρνούμαστε, ποτέ δεν απορρίπτουμε τέτοια αιτήματα, πάντοτε προσπαθούμε να βοηθούμε τους συναδέλφους που μας ζητάνε τη βοήθειά μας, ε, οπότε οι υποθέσει τρομοκρατία είναι σίγουρα μέσα στι υποθέσεις όπου έχουμε λάβει αιτήματα ε, για συνδρομή. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σας πω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διασύνδεση ανάμεσα στη μετανάστευση και την τρομοκρατία ή ότι έχουμε περισσότερες επιθέσεις, ε, υποθέσεις μάλλον λόγω μετανάστευση. Υπάρχουν πολλέ ερμηνείε εξηγήσεις που μπορεί κανεί να δώσει γιατί έχουμε περισσότερε τρομοκρατικέ υποθέσει θα, μπορούσε, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και οι αντιτρομοκρατικές αρχές ε, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι παλιότερα σε εμά και γι' αυτό και μα δίνουν περισσότερε υποθέσει, μα ζητούν περισσότερε πληροφορίε. Για το αντιτρομοκρατικό μητρό, πρέπει να σα πω ότι δεν ανακαλύψαμε ε, τίποτα από την ε, αρχή, δεν βασιστήκαμε σε κάποιο νέο νομικό μέσο. Ε, βασιζόμαστε πάντοτε στην ε, απόφαση Συμβουλίου 671 ε, του 2005 του Συμβουλίου, ξαναλέω, για την ανταλλαγή υποθέσεων στις τρομοκρατικές υποθέσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε στις χώρες ε, ρεαλιστικές λύσεις οι οποίες θα τις βοηθούν να μας στέλνουν αυτού του είδους τις πληροφορίες δεν είναι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι, δεν είναι βάση δεδομένων με μυστικές πληροφορίες εμείς ε, συλλέγουμε μόνο πληροφορίες για ε, ποινικέ διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αν υπάρχουν δηλαδή δικαστικές διερευνήσεις υποθέσεων, αν υπάρχουν ε, καταδίκες δηλαδή. Αυτό είναι ο στόχος και ο στόχος είναι πάντοτε να διασυνδέουμε αυτές τις, δύο, αυτές τις διάφορες υποθέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη, όπως εξήγησα και εισηγητικά στην παρουσίασή μου. Νομίζω ότι υπήρχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Τι κάνουμε. Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων έχει διάφορα, διάφορες φάσεις. Πρώτον πρέπει κανείς να προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία. Μετά πρέπει να τα παγώσει, να περάσει στην κατάσχεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Ε, υπάρχουν διάφορα στάδια λοιπόν. Η Eurojust βοηθά σε, αυτά, σε όλα αυτά τα στάδια, σε όλες αυτές τις φάσεις. Ε, με διαφορετικούς τρόπους γιατί σε κάθε στάδιο χρειάζεται διαφορετικό είδος ε, βοήθειας. Όταν υπάρχουν αποφάσεις κατάσχεσης εμείς εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι κατασχέσεις μπορούν πράγματι να γίνουν ε, στη χώρα όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία, διότι ξέρετε ότι σε διάφορες χώρες μπορεί να συντρέχουν ή να ισχύουν διάφορες προϋποθέσεις για να περάσει κανείς σε κατάσχεση. Υπάρχουν και διάφοροι σκοποί βεβαίω που συνοδεύουν την κατάσχεση. Κάποιες, κάποιες φορές γίνεται κατάσχεση χρημάτων για την αποζημίωση θυμάτων, κάποιες φορές ε, ε, πρέπει ενδεχομένως να κάνεις μια κατάσχεση χρημάτων ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά ως αποδεικτικό στοιχεία σε μια ποινική διαδικασία. Κάποιες φορές αποτελούν και αποδεικτικά στοιχεία ε, ε, στην, στο πλαίσιο της διερεύνησης κάποιας ποινική υπόθεσης. Οπότε υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις αν θέλετε. Εμείς πάντοτε παρέχουμε ε, συμβουλές προς τις χώρες για το πώς μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση ώστε να τις βοηθήσουμε να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους για να γίνει η κατάσχεση ε, στην χώρα στην οποία βρίσκονται τα περιοσιακά στοιχεία. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει, πρέπει να σας πω ότι εδώ πράγματι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, και όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε, για να δούμε ακριβώς τι έχουμε κάνει. Στο παρελθόν, ε, με μεγάλη περηφάνεια, ε, ε, μετρούσαμε, αν θέλετε, την, τις επιδόσεις μας σε, μια σειρά από τομείς όσον αφορά τον αριθμό των, των μελών των ομάδων διερεύνησης σε διάφορους υποτομείς, αν θέλετε, της ποινική δικαιοσύνης και μιλώντας μαζί σας έχουμε καταλάβει ότι δεν αρκούν όλα αυτά. Θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα, θέλετε συγκεκριμένα ποσά που έχουν κατασχεθεί ε, και αυτό ε, είναι μια δουλειά την οποία την έχουμε ξεκινήσει. Την ξεκινήσαμε για παράδειγμα στην Ουγγαρία όπου ε, σε συνεργασία με τις Ουγγρικές εισαγγελικέ Αρχές καταφέραμε και προσδιορίσαμε πόσα ακριβώς ήταν τα χρήματα που ε, αφορούσαν οι υποθέσεις που είχαν παραπεμφθεί στην ε, Eurojust. 40 ε, εκατομμύρια, μπορώ να σας δώσω αυτό το στοιχείο, 40 εκατομμύρια ήταν οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών που έγιναν στην Ουγγαρία. Αυτό είναι άλλωστε και ο προπολογισμό, αν θέλετε, της τη ίδια τη Eurojust. Και όλα αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στα κράτη-μέλη. Εμεί ω Eurojust δεν κρατάμε ούτε ένα ευρώ. Οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα ε, ένα αποδεικτικό στοιχείο, αν θέλετε, για το πώς η Eurojust βοηθά τα κράτη-μέλη και τις αρχές τους. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπήρξε και ένα ερώτημα για, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το EPPO. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς προσβλέπουμε πραγματικά στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε πλέον έναν εταίρο με τον οποίο θα μπορούμε να, να ε, μιλήσουμε για μια συμφωνία συνεργασίας και νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα, θα μας φορτώσει με ακόμα περισσότερη δουλειά ε, θα μας παραπέμπει πολλές ε, υποθέσεις και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού για να καθοριστούν οι αρμοδιότητες, ποιος θα κάνει τι. Ξέρετε ότι πέντε χώρες δεν συμμετέχουν στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε εξακολουθούμε εμείς να έχουμε την αρμοδιότητα για αυτές τις χώρες. Θα δημιουργηθούν ε, κάποια ε, προβλήματα όσον αφορά το πώς θα συνεργαστούμε. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν διάβλη επικοινωνίες, επικοινωνίας, ε, ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στις διάφορες βάσεις δεδομένων και όπως είπα περιμένουμε να έχουμε αύξηση ε, του αριθμού των υποθέσεων και από τρίτες χώρες και Brexit τέλος γιατί και αυτό ήταν πολύ σημαντικό ερώτημα. Είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους μας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν γίνει εκτεταμένες συζητήσεις, έχουμε ε, διάφορα σενάρια και περιμένουμε το πολιτικό αποτέλεσμα της όλης αυτής ε, διαδικασίας. Πάντως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όποιο και αν είναι το σενάριο που θα επαληθευτεί, έχουμε ε, ήδη εγκρίνει και θεσπίσει τα μέτρα και θα εξασφαλιστεί η συνεργασία και μετά το Brexit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για την προσπάθεια που καταβάλατε να μας βοηθήσετε για να μην ξεφύγουμε και από το χρονικό πλαίσιο. Γιατί φυσικά είναι σημαντικά τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη να... Ε, και τις τελευταίες ε, παρατηρήσεις που έγιναν για, το, για την ΕΠΟ ότι το άρθρο 86, σύμφωνα με το άρθρο 86, η ΕΠΟ θα πρέπει να την διαχειριστεί η Eurojust. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσουμε πάρα αυτά στο επόμενο θέμα της ημερησίας διαταξής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολουθήσεις για τα Ναρκωτικά. Έχουμε τον επικεφαλής ε, Τη υπηρεσία εδώ, στην αίθουσα ήδη. Όπω σα time Όπως σας είπα, ξεπεράσαμε το χρονικό όριο και φυσικά είχαμε πολλά να πούμε. Δεν ε, θέλω να σας καθυστερήσω λοιπόν και να περάσουμε στην επόμενη, στο επόμενο κέντρο. στο σύνολο αυτών των κέντρων που εξετάζουμε. Ευρωπαϊκό Κέντρο λοιπόν παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας. Έχουμε τον επικεφαλή λοιπόν της Υπηρεσία αυτής που έχει έδρα στη Λισαβόνα και θα μας κάνει μία εισαγωγή για το έργο της ε, υπηρεσία, ε, του κέντρου. Κυρίως επικεντρωνόμενος ε, στο 2018 και 2019. Έχετε 10-15 λεπτά στη διάθεσή σας και μετά θα ακολουθήσει ο συνήθις γύρος ε, έρωτα Σάνα. Όσοι θέλετε λοιπόν να κάνετε ερωτήσεις, σχόλια. Παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Γιατί έχουμε και άλλα κέντρα να εξετάσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι βουλευτέ Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και πάλι ενώπιόν σας. Κάποιου από εσά σας γνωρίζω για πρώτη φορά, κάποιου άλλου σα έχω ξανασυναντήσει. Είναι η πρώτη συναντρίαση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όπως σας είπα, εν συντομία θα σας κάνω μία παρουσίαση και θα, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας για τις δραστηριότητε μα σε ό,τι αφορά το που βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Να σας υπενθυμίσω ότι οι πού ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε για την τοξικομανία και τα ναρκωτικά. Αρχές δεκαετίας του 80, 80 επιδημίες οι οποίες ε, διαδοθήκαν σε όλη την Ευρώπη και σκότωναν ε, τεράστιο ρυθμό ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες επιδημίες ε, επιδεινώθηκαν με την εμφάνιση του HIV, του ΕΠΣΗ και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την Προεδρία του Φρανσουά Μιτερά με επιστολή του 89 προς τα άλλα κρατημέλη αποφάσισε να αντιεξαγάγει μια μελέτη εφικτότητας για να διαπιστώσει κατά πόσον χρειάζεται και πώς θα λειτουργούσε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την τοξικομανία. Γι' αυτό λοιπόν έτσι ξεκινήσαμε τις δευτεριότητές μας. Ο κανονισμός εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 1993 ξεκινήσαμε να λειτουργούμε στη Λισαβόνα τον Ιανουάριο του 1995. Άρα του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 25 μας χρόνια. 25 χρόνια παρακολούθησης και εποπτείας. Ποια είναι λοιπόν η προσταθέμενη αξία μας. Συμβάλλουμε για μια πιο ασφαλή και πιο ασφαλή και υγιή Ευρώπη με πολιτικές και δράσεις. Έχουμε δύο πυλώνες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι αυτό αποτυπώνει και τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα ναρκωτικά. Βασιζόμαστε κυρίω σε δύο άρθρα τη συνθήκη, δικαστική συνεργασία και για την ε, δημόσια υγεία. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν δύο τέτοιε ομάδε δραστηριοτήτων με συγκεκριμένου ε, στρατηγικού στόχους και συμβάλλουμε και στην εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια υγεία, έγκυρη προειδοποίηση κτλ. και στον τομέα της ασφάλειας για τους ανθρώπους που μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα χρησιμοποιήσω και μία λέξη η οποία δεν είναι και πολύ μοναδική, ιδιαίτερη, γιατί το σύστημα το οποίο έχουμε στην Ευρώπη είναι μοναδικό. Το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τις ε, νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Το σύστημα το πρώτο ήρθε το 1997 με την πρώτη κοινή δράση, η οποία αποφασίστηκε λόγω το, της εμφάνισης των νέων συμφετικών αυτών ναρκωτικών που εμφανίστηκαν σε κάποια κρατημέλη και σε κάποια κρατημέλη ήδη ε, σκότωναν ε, τους, κάποιους από τους πιο νέους μας πολίτες. Το σύστημα αυτό λοιπόν ήταν μοναδικό γιατί υπάρχει ε, ένα νέο τέτοιο σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας έχει 30 μέλη. Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Τουρκία. Και ουσιαστικά συμπληρώνουμε το έργο των ε, εθνικών ε, παρατηρίων 28 κράτη-μέλη και Νορβηγία και Τουρκία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια ως υποψήφιες χώρες. Τώρα επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και με άλλες χώρες. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Γιατί είναι μοναδικό λοιπόν το σύστημα, γιατί. Βάζεις ένα μοναδικό πλαίσιο δεδομένα που καλύπτουν και την εφαρμογή του νόμου και τις, τα περιστατικά, τα θέματα δημόσιας υγείας, τα θέματα τοξικομανίας. Αυτό λοιπόν είναι μοναδικό Έτσι λοιπόν να εντοπίζουμε τα προβλήματα που αναδύονται σε πρώιμη φάση. Υπάρχει μία σύντομη περίοδος ε, αξιολόγησης και στο τέλος αυτής της εξάμενης περίοδου τα κρατημέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για να τεθεί μία ουσία υπό έλεγχο, το οποίο παίρνει έξι μήνες έως 2-3 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτό το μοναδικό εργαλείο. Επίσης, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο όταν μπαίνει υπό έλεγχο μια ουσία είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ε, δεδομένα τα οποία συλλέγονται σε επίπεδο κρατούς μέλους συνενώνοντας στοιχεία και των αστυνομικών δυνάμεων και των ε, δυνάμεων επιβολή νόμου, σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Κάποια προϊόντα λοιπόν στον τομέα της δημόσιας υγείας. Προφανώς υποστηρίζουμε όλες ε, τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί και τα πρότυπα βέλτιστης ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατα θα προσέξετε ότι κάναμε μία μία δημοσίευση για την ιατρική χρήση της κάναβης και υπάρχει πλέον ένα ξεχαριστό εργαλείο για τη χρήση της κάναβης. Θα το θίξω το θέμα αυτό σε λίγο. κοιτώντα όλες τις συμβολές μας στον τομέα της ε, υγείας, της δημόσιας υγείας, προφανώς ε, συνεργαζόμαστε με τις αρχές ε, των Υπουργείων Εσωτερικών και με τη Eurojust και με τη Europol όπως είπε και ο προηγούμενος μελτής. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με την Europol, είμαστε σε στενή συνεργασία για την αξιολόγηση των απειλών, αλλά και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχεδίων δράση. Γιατί, όπω θα ξέρετε, υπάρχουν προτεραιότητε. Πολλέ προτεραιότητε, λοιπόν, αφορούν ναρκωτικά. Παρακολουθούμε και αναλύουμε τα ναρκωτικά, το Darknet, και πριν από ένα χρόνο κάναμε με τη σχετική δημοσίευση με την ε, πλήρη ιστορία και εξέλιξη κάποιων σκοτεινών τέτοιων δικτύων που πολλούν ναρκωτικά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά συμβάλλουμε και στον ε, κύκλο της αστυνομία για την ανάλυση των στοιχείων αυτών. Κάθε τρία χρόνια, 3 Δεκεμβρίου, θα δημοσιευτεί η έκθεσή μας για την αγορά ναρκωτικών μαζί με την Europol. Αυτές είναι λοιπόν ως συντομία οι δημοσιεύσεις μας και τα προϊόντα μας. Επίση, επικεντρωνόμαστε στην εξωτερική διάσταση τη ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Προεδρία του Συμβουλίου για τα Ναρκωτικά, τι διμερεί διαλόγου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του περιφερειακού διαλόγου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, υποστηρίζουμε και συμβάλλουμε και στα περιφερειακά προγράμματα για τα ναρκωτικά όπως το Κόπολα, το οποίο είναι ένα πολύ καινοτόμο σύστημα το οποίο ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και πλέον συνδυάζει και τις χώρες της Καραϊβικής. Έχουμε και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και πρόσφατα και ένα νέο πρόγραμμα με τη χρηματοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις γειτονικές χώρες. Αυτά ε, ε, εντάχει ε, αυτό είναι ένα πανόραμα των δραστηριοτήτων μας. Μου ζητήθηκε τώρα να σας παρουσιάσω ε, εν συντομία το πώς έχει η κατάσταση για τα ναρκωτικά. Γιατί εξακολουθούμε να ανησυχούμε για τα ναρκωτικά. Έχουμε πρόβλημα με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη σήμερα. Το ερώτημα αυτό μπορεί να μην είναι τόσο πρόφανες για όλους μας, για τον απλό λόγο ότι όταν αποφασίστηκε να υπάρξει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά, όταν κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει Ευρωπαϊκή Στρατηγικά για τα Ναρκωτικά, ήταν επειδή ο κόσμος πέτσανε στις μεγάλες πόλεις, στους δρόμους. Και χάρη στις προσπάθειες των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πλέον ευτυχώς δεν το παρατηρούμε πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν έκαναν επενδύσει όλα τα κράτη-μέλη, γι' αυτό υπήρξε υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τοξικομανία και Ανακριτικών και των άλλων ευρωπαϊκών υπηρεσιών για τον εντοπισμό των τέτοιων κρουσμάτων. Πώ έχει λοιπόν η κατάσταση σήμερα, κοιτώντα τι εξελίξει των τελευταίων χρόνων και συναντήθηκα με την ε, βελγική αστυνομία σήμερα. Να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια της προσφοράς όλων των ουσιών, όχι μόνο της κοκαίνης, γιατί θα ακούσετε πολλά για την κοκαίνη το Δεκέμβριο στην έκθεσή μας, αλλά και της ηρωίνης των οπιοειδών. Χτες, μάλιστα, είχε ένα άρθρο ε, η Guardian, την οποία, το οποίο επιβεβαίωσε η βελγική αστυνομία 1,2 τόνοι αμα, ηρωίνης που κατασχέθηκαν από την ε, αστυνομία της Βρετανίας και της Ολλανδίας. Και έχουμε και άλλα ναρκωτικά που έρχονται στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάτε επίσης μία μεγάλη διαφορά σε σχέση με πριν από 30 χρόνια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι μεγάλος παραγωγός κάναβης, ε, ε, συμφετικών ναρκωτικών, έκσταση, μετα, με MDMA, μεταμφεταμινών και να σας πω ότι στις ε, χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι τεράστιο το πρόβλημα με τις μεταμφεταμίνες. Στην, Ευσφαλή, στην Αυστραλία επίσης ε, τεράστιο το πρόβλημα και στη Νέα Ζηλανδία. Και αν ένα πράγμα ευχόμαστε είναι να μην μας χτυπήσει η, η ίδια επιδημία, γιατί πραγματικά έχει τραγικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών. Δεύτερη παρατηρήση. Τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τη σύσθεση των ε, ναρκωτικών. Το 2000, να σας πω, είχαμε 65 μιλιγκράμμα και έκσταση σε κάθε εμ, χάπι έκσταση. Σήμερα ένα μέσο χάπι έκσταση έχει 180 μιλιγκράμμ δραστικής ουσίας ε, και κατά το όριο 240 έως και 310 μιλιγκράμμ. Και αυτά τα βρίσκουμε με, τις, τα μηχανήματα ελέγχου της α, ε, σύνθεσης των χαπιών αυτών. Αυτό που δεν ε, βλέπουμε ευτυχώς ακόμα είναι τεράστια αύξηση της κατανάλωσης. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει. Οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν καμία. Ε, πέρα από το MDMA τύπου έκσταση. Σήμερα Πέρσι εντοπίστηκαν 55 ε, νέες ουσίες. Μία κάθε εβδομάδα. Παλιά ήταν και δύο την εβδομάδα. Πέρσι λοιπόν από το σύνολο των 720 ουσιών που εξακολουθούμε να παρακολουθούμε, 320 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά πέρσι και έχουμε και δύο ε, Ουσίε που ετέθησαν υπό έλεγχο μετά από απόφαση του Συμβουλίου για αξιολόγηση κινδύνου. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά του θανάτου που προκαλούνται από τα ναρκωτικά. Και το προηγούμενο Σάββατο δημοσιεύθηκαν ε, σχετικά στοιχεία για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκριση για το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα αυτό. Καταρχά, αυξάνεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ωστόσο, έχουμε περίπου 9.500 θανάτους με 10.000 θανάτους ε, κάθε χρόνο στο, στη ΣΥΠΑ. Οι θάνατοι αυτοί είναι 72.000. Το ίμιση εξ αυτών από αμφεταμίνες ε, στη ΣΥΠΑ. Αυτή η επιδημία λοιπόν δεν είναι η ίδια όπως το παρελθόν, αλλά βλέπουμε να εμφανίζονται νέες ε, ουσίες να εμφανίζονται. Ήδη φέτος έχουμε σημειώσει 40 νέες ουσίες που έχουν εμφανιστεί και κάποιες από αυτές από μια νέα οικογένεια την οποία δεν ε, παρακολουθούσαμε στο παρελθόν. Είναι πολλές οι προκλήσεις και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις επενδύσεις, αλλά να προσαρμόσουμε και την απάντησή μας στις προκλήσεις αυτές. Αυτή είναι μία πρώτη πρόκληση. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω όλες τις προκλήσεις που έχουμε, δεν έχουμε χρόνο για σήμερα, αλλά μία άλλη πρόκληση είναι οι αλλαγές στην αριθμιστική πολιτική σε ό,τι αφορά την κάναβη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει αυτό και αλλάζει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ιατρική χρήση της κάναβης και των καναβοειδών και σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση της κάναβης. Ακόμα και το γεγονός ότι αλλάζει τόσο πολύ κατάσταση σε διάφορες πολιτείες της Ευρωπα... των ΗΠΑ έχει αντίκτυπο και θα έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς υποτίθεται ότι σας ενημερώνουμε, σας δίνουμε επιστημονικά στοιχεία για να μπορείτε να καταλαβαίνετε και να παρακολουθείτε την κατάσταση. Για να κλείσω, μου, ζήτησε, ζητήθηκε να πω δύο λόγια για το ποια είναι η απόδοσή μας και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Για την επίδοσή μας. Να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος γιατί τουλάχιστον από τότε που είμαι επικεφαλής του κέντρου, καταφέραμε να δίνουμε καλύτερες υπηρεσίες ε, για τα χρήματα που ξοδεύουμε. Έχουμε 98,02% εκτέλεση πληρωμών. Ρεκόρ για ένα τέτοιο κέντρο. Και είναι το τρίτο ετός ε, που έχουμε τέτοιο επίπεδο ανταπόκριση στις δεσμεύσεις μας. Άρα, εγώ δεσμεύομαι ότι πρώτα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε όσο πιο καλά γίνεται τους πόρους που έχουμε και μετά θα κοιτάξουμε. Επίσης, ε, μία επιπλέον αξιολόγηση έγινε πέρσι και λάβαμε ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απόδοσή μας είναι εξαιρετική. Να σας πω ότι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί η αξιολόγηση κάλυψε τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τμήμα της ε, θητείας του προκατόχου μου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δείκτες για την απόδοσή μας καταδεικνύουν ότι είχαμε την καλύτερη αξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση ως τώρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα ή άσπρα και προφανώς υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Ε, κάποια, μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η χρηματοδότηση δεν ε, είναι πολύ πρωτοτυπό αυτό. Πολλά ε, κέντρα το έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουμε το θέμα των ε, δαπανών για τους μισθούς των υπαλλήλων, που είναι 70% των εξόδων μας. Έχουμε επενδύσει καταρχάς σε κτίρια, μάλλον συγγνώμη, σε επένδυση στη δημιουργία δυναμικού που έλειπε και φέτος αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τις, ε, κατά 1,3 εκατομμύρια τις δαπάνες μας. Κατά δεύτερον, έχουμε το πρόβλημα που ανέφεραν όλοι οι συνάδελφοί μας. Αν συνεχίσουμε να αυξάνουμε αυτά τα αρχικά σενάρια, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φτάσει η χρηματοδότηση για το κέντρο μας. Αλλά από τότε που συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε να πούμε ότι η Επιτροπή σα πάντα μα έδινε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και με την νέα αυτή Επιτροπή θα συνεχίσετε να κάνετε διαφορά για μα. κύριε Χορστέλ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ολοκληρωμένη η παρουσίασή σα όσον αφορά το κέντρο παρακολούθηση και επίση έτσι φάνηκε το πώ ε, συνδέονται τα επιμερου ε, ζητήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά από την άλλη μεριά έχουν ε, πολιτική σημασία. Και το έχουμε αναφέρει, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Ναι, ακριβώς όλα αυτά τα περίπλοκα προϊόντα και ναρκωτικά τα ε, οποία γνωρίζουν όλο και περισσότερη ζήτηση και είναι μια πρόκληση για την πολιτική μας όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Τώρα πήγε ο χρόνος, αλλά να βρούμε χρόνο για τους ανθρώπους που να λάβουν το λόγο. Βλέπω οι, όποιοι επισμενιστές είναι εδώ ότι θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να μιλήσουν. Κυρία Σάντος, κυρία Κελέα τρίτος, ο Γιώργος Πακατσίνη και ένας άλλος συνάδελφος. Θέλετε και εσείς το λόγο, κυρία. Μάλιστα. Ναι, ναι, λέει η κυρία Σάντος. Οπότε εσείς μιλήστε πρώτοι και στη συνέχεια να καλύψουμε όλους όσους ζήτησαν το λόγο. Αλλά παρακαλώ, παρακαλώ. Ε, όσο μπορείτε πιο συγκεκριμένοι, σύντομοι, μονόλεπτες ερωτήσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, θα υποβάλω χωρίς πολλά πολλά την ερώτηση. Να στα πω ή στα πορτογαλικά. Και έτσι με τη μετάφραση θα καταλάβετε όλο όσα αλλιώς. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για το έργο σας. Γιατί ε, ε, αυτό κάνει τη διαφορά όσον αφορά και τον ε, τομέα της δημόσιας υγείας από την αρχή της διαδρομής της αυτή η υπηρεσία έχει κάνει την ε, διάφορα και ήταν εντυπωσιακή η βελτίωση ε, των όσων ε, κάνουμε για τους πολίτες. Οπότε, μπράβο σας και πάλι τώρα. Για να δούμε τι γίνεται με το dark net, το, το, το, το σκοτεινό κομμάτι του διαδικτύου. Τα πράγματα εκεί είναι οίκιστα, ε, διαφανή. Οπότε θα πρέπει κανένας να πασχίσει και να καταλάβει πώς λειτουργεί η αγορά σε αυτό το κομμάτι το σκοτεινό του διαδικτύου. Πρώτα και ολόκληρο αγώνα που πρέπει να κάνω σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Κέλλερ, για την συγκριτή σα. Έχω πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Δύο συγκεκριμένε, λοιπόν. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την ε, αστυνομία. Όταν ε, κάνει κάποιε επιχειρήσει, ε, ανακτά, κατάσχει κάποιες ποσότητες ναρκωτικών, μεγάλες και μικρές. Υπάρχουν επομένως ε, για κάποιες περιπτώσεις που έχουμε μικρές ποσότητες που κατάσχονται και υπάρχει ζήτημα για στο πώς διατίθενται αυτές οι μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Τι τις κάνουνε. Πώς θα αποφύγουμε το να μην πάνε στο περιβάλλον αυτά τα ναρκωτικά και υπάρχει θέμα και ιδιαίτερα με την, ε, με Επομένω, πρέπει κανεί να διεκπεριώσει το θέμα για να μην υπάρξει κάποιο είδου υπεξαίρεση αυτών, αλλά για την άλλη να μην πάνε όπω όπω το περιβάλλον έτσι χωρί κάποια επεξεργασία. Άλλη ερώτηση. Κάνετε κάποιε εκστρατείε ε, ε, χαρακτήρα πρόληψη, συγγνώμη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε αναλύσει που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι έφηβοι, κάποιοι νέοι που παίρνουν ναρκωτικά. Ε, αυτό το shit ε, και ε, οδηγούνται σε κάποιο τους ε, ψυχιατρικές ε, παθήσεις. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη ως γνώση. Όλα αυτά τα, τα λαμβάνετε υπόψη για την στρατηγική, την πολιτική σας για νομιμοποίηση της κάναβης κύριε Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτης δεν λέγεστε. Αρβανί... Κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήταν πληρέστατη. Θέλω να σας πω ότι εγώ σας γνωρίζω, εσείς δεν με γνωρίζετε. 30 χρόνια ασχολούμαι με, την, με το θέμα της φύσης και της εξάρτησης ναρκωτικών ουσιών. Α, ως αντιπρόεδρος στις θεραπευτικές κοινότητες της Ελλάδας, το ΚΕΘΕΑ. Και μέλος... Ε, μία επισήμανση θέλω να κάνω, δεν είναι καν ερώτηση. Δεν είναι μόνο η αγορά η οποία πρέπει να μας απασχολεί στο θέμα της χρήσης, της εξάρτησης και του θανάτου των ανθρώπων από τις ουσίες. Είναι και η ανάγκη των ανθρώπων σε εισαγωγικά που πάνε στη χρήση. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να επισημάνω και να καλέσω τους συναδέλφους μου, όλους τους συναδέλφους από όλες τις δημοκρατικές πτέρυγες και κόμματα. Να στηρίξουν την ε, δουλειά σας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν 16 ε, εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, 266.000 περίπου. Το Συμβούλιο πρότεινε μείωση. Διαφωνούμε πλήρω ω Γκουέ και ω αριστερά και εγώ προσωπικά με αυτό το πράγμα. Είναι εγκληματικό δηλαδή να λέμε ότι από τη μία μπράβο στο έργο σα και από την άλλη σα κόβουμε αυτό που έχουμε ανάγκη σαν πολίτε. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι πολίτε, άνθρωποι, παιδιά που χάνονται καθημερινά στι γειτονιέ μα στην Ευρώπη. Και προτείνουμε, και κλείνω με αυτό. Καταθέσαμε στην ΚΟΕ, εμεί από την ΚΟΕ και εγώ και ο σύντροφο Κόκαλη, την τροπολογία 5803. Προτείνουμε την αύξηση του ποσού στα 17.839.000. Σας εκλυπαρώ και σας κάνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους, στους γονείς, επειδή έχω ζήσει αυτή την ιστορία και τον πόνο των ανθρώπων, σε αυτό το θέμα να μην κάνουμε πίσω. Εδώ η Ευρώπη μπορεί να δείξει πραγματικά το πρόσωπό της και την αλληλεγγύη Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το χρόνο που έφαγα. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Ποκατσίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε για την εισήγηση. Έχω την εξή ερώτηση. Δεδομένου ότι ο νόμος ε, σε σχέση με την χρήση της τραπευτικής κάνοβης ε, ποικίλουν, ποικίλουν πάρα πολύ από τη μια χώρα στην άλλη, στην Ένωση. Τι λέτε για την ε, πρωτοβουλία της Φιλανδικής Προεδρίας όσον αφορά ε, τον ορισμό μιας κοινή ευρωπαϊκής θέσης όσον αφορά τις ε, συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, όσον αφορά την θεραπευτική κανοβική της συναφής ουσίας. Mr. Garand. Γαρό. Γαρό, γαρό. Γαρό, ονομάζομαι. Α, συγγνώμη. Συμπαθάτε με το πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση και συνέφεια μεταξύ αύξησης εγκληματικότητας και αύξησης κατανάλωσης ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά ε, οδηγούν σε λάθρεμπόριο, σε εγκληματικότητα ε, που δεν είναι συνδυόμενα άμεσα ε, με τα ναρκωτικά όπως το διακίνηση ναρκωτικών αλλά όλα αυτά είναι εγκλήματα και μας τα είπατε κι εσείς έξω από τα δόντια και υπάρχει αύξηση αισθητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω με αυτά τα νέα ναρκωτικά, τα νέα προϊόντα. Οπότε, σε συνέχεια των όσων είπατε, σε συνέχεια των επαφών σας με άλλες υπηρεσίες, υπάρχει και αύξηση ε, της εγκληματικότητας στην Ένωση. Μπορείτε κάτι να κάνετε κάτι παραπάνω από τις ε, πολιτικές που υπάρχουν στην Ένωση, τις ε, κατασταλτικές πολιτικές σε σχέση με τα ναρκωτικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα μπορούμε να αποσπάσουμε ε, για όλα αυτά τα εγκλήματα. Κύριε Μπρικμόντ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον έχετε και κάποιους κριτήρια για το ποια κράτη έχουν πιο αποτελεσματική νομοθεσία όσον αφορά την ποινικοποίηση των πράξεων των ε, ναρκωμανών, τι γίνεται με την κάλυψή τους από τις ε, πολιτικές υγείας κλπ. Και ποιο είναι το κόστος. Και Ακούσαμε ε, τις ερωτήσεις, πάλι έχουμε περιβεί το χρονικό όριο. Έχετε τώρα τη σκητάλη για να καλύψετε όλες αυτές τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχετε το λόγο. Και Χόστελ. Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Λέει στα γαλλικά και στα πορτογαλικά. Πρώτα-πρώτα για την ερώτησή σας για το σκοτεινό δίκτυο, το Darknet. Ναι, είναι σημαντικό να αναδείξουμε το ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι του διαδικτύου. Συνεργαζόμαστε με την Europol, υπάρχει ένα κέντρο παρακολούθησης και παρακολουθούμε τι γίνεται με το έγκλημα και υπάρχει στενή συνεργασία του παρατηρητήου και της ε, Europol. Γίνεται στρατηγική ανάλυση των δεδομένων και προχωρούμε, προσπαθούμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Δεν είναι τόσο μεγάλη και η δραστηριότητα σας στην αγορά των ναρκωτικών, αλλά συνεχώς εντείνεται και αυξάνεται. Πάντως, από ό,τι φαίνεται είναι περιορισμένη η εμβέλεια του Darknet όσον αφορά τη διακίνηση των ναρκωτικών. Δεν είναι δουλειά μας να επέμβουμε, να παρέμβουμε σε αυτό το επίπεδο. Ε, ε, αυτό είναι δουλειά της Europol και των κρατών μελών. Ε, βέβαια και θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Darknet και γενικότερα στο διαδικτύο. Και όλα αυτά να τα καλύψουμε και στην έκθεσή μας που θα δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Οπότε όπου τα θέλετε που είσαστε προσκεκλημένοι μας ή στην Ελισσαβόνα για να τα πούμε από κοντά. Ε, κύριε Κελεδρό, όσον αφορά τις κατασχέσεις ναρκωτικών υπάρχουν ε, διατάξεις που δεν γνωρίζω, ε, δεν είμαι αστυνομικός υπάλληλο, οπότε σε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας δεν κάνω τίποτα, αλλά υπάρχουν σαφείς οδηγίες και διατάξεις στα κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή τους, ε, εντάξει, βέβαια. Πολλέ φορέ δεν υπάρχουν καν διατάξει πρέπει να τις θεσπίσει κανεί και κατόπιν θα πρέπει κανεί να τις ε, τηρεί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αυτό το οποίο κάνουμε και με την ευκαιρία ε, να σας ενημερώσω όλους σχετικά, είναι ότι αναλάβουμε την αρμοδιότητα με την Europol ε, για να δούμε τι γίνεται με τα στατιστικά δεδομένα, τους δείκτες όσον αφορά την προμήθεια ε, και βλέπουμε στις κατασχέσεις τι γίνεται με την καθαρότητα του προϊόντος. Έχουμε νέα νηματολογία και νέες κατηγορίες προϊόντων που τώρα έχουν σχέση με τις κατασχέσεις. Οπότε και σε εθνικό επίπεδο, όπως είπε ο Βέλγος συνάδελφος, υπάρχει ένα σχέδιο ούτως ώστε να υπάρξει πληροφόρηση όλων για το τι γίνεται και να υπάρχει κάποιο είδους κεντρική διαχείριση των πληροφοριών. Βέβαια κάθε χώρα έχει διαφορετική παράδοση, ε, διαφορετική διεκπαιρέωση και το θέμα είναι βέβαια να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Οπότε καταβάλλεται προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση τώρα μας είπατε και για το περιβάλλον, όλα αυτά θα τα πούμε στην έκθεση του Δεκεμβρίου, διότι βεβαίω και το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αυτό που μας ε, τονίσατε, το τι κάνει κανείς με τις κατασχεθήσεις ποσότητες. Είναι μεγάλο περιβαλλοντικό το πρόγραμμα. Αυτό και συνέβη και με την παραγωγή των νησιών. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη. Όχι, δεν κάνουμε ε, εκστρατείε πολιτικού χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι δουλειά μας ε, και εσεί αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε την εντολή και να την πάτε προ αυτή την κατεύθυνση. όμω στην Ευρώπη εδώ και δέκα χρόνια έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης. Συγγνώμη, την είχαμε, την είχαμε στο παρελθόν. Αλλά, αλλά ε, δυστυχώς αυτή η εβδομάδα που είχε καθιερωθεί ε, καταργήθηκε. Δεν ξέρω, μακάρι να ξαναξεκινήσει αυτή η ενημερωτική καμπάνια. Οπότε εμεί προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να καταγράψουμε, να συνεργαστούμε με όλους τους εμπειρογνώμους των κρατών για τις ε, καλές πρακτικές για να μειωθεί η ζήτηση. Να, αυτό έχει σχέση με τη μείωση του κινδύνου, με την πρόληψη, οπότε η προτεραιότητά μας στις στρατηγικές μας είναι να μπορέσουμε όλα και περισσότερο να συνεργαστούμε για να εφαρμοστούν ε, προγράμματα πρόληψης στα κρατη Και πάμε καλά, έχουμε πάρα πολλά προγράμματα. Ε, καλά τα δέχονται οι νέοι. Βέβαια, πολλές φορέ είναι ξεπερασμένα τα προγράμματα και πολλέ φορέ έχουν και τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Οπότε έχουμε και τον Ευρωπαϊκό ε, Οδηγό όσον αφορά τις ε, παρεμβάσει κοινωνικού υγειονομικού χαρακτήρα και σύντομα θα έχουμε ένα νέο κύμα ε, με νέα μέσα πολιτικής. Ραντεβού τον Οκτώβριο στην Λισαβόνα έχουμε με τις Πορτογαλικές αρχές μια ε, διοργάνωσε μια πολύ μεγάλη, πιο μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση όσον αφορά ε, κάθε είδους τοξικομανία για την Ευρώπη. Τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Θα σας στείλω τα σχετικά. Θα διαβάσουμε στη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ. Κύριε Αρβανίτη. Άλλος, θα έχουμε το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες, οπότε θα το συζητήσουμε Πάλι μια φορά σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Yeah. Next one. Um, Επόμενος. Άλλη ερώτηση αφορούσε τον Ιταλό συνάδελφο για την ε, Κάναβη. Θα μπορούσα να στα πω Ιταλικά, αλλά θα ζοριστώ περισσότερο, θα περιοριστώ στα Αγγλικά. Αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή πρώτα-πρώτα εμεί στο παρατηρητήριο δεν ε, καλύπτουμε την ε, θεραπευτική κάναβη. Γιατί αν πάμε στην ιατρική και στη φαρμακολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και στο Baobab ε, και στο φοινικό δέντρο. Όμως, η βασικό συστατικό είναι για μας το να μιλήσουμε για τα αποστάγματα, τη, την πικροτροπική κάναβη κλπ. Για την κάναβη, για την κάναβη. Ε, και αναφέρατε την φιλανδική πρωτοβουλία και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο στόχο είναι πάρα πολύ σωστά ταγμένο. Όμω αυτό είναι συνέχεια τη κοινή προσπάθεια των κρατών μελών, ούτω ώστε να υπάρχει σε επίπεδο ΟΗΕ ενιαία τοποθέτηση. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τις καινούργιες χώρες και κάποιες άλλες χώρες. Ε, αυτό είναι πρόκληση και για μας, τις υπηρεσίες, οργανισμούς, γιατί υπήρξε πρόταση του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι σοβαρός οργανισμός και άπαξ και λένε ότι η κάναβη ή κάποια από τα στατικά της θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, διαφορετικά. Δεν το λένε από ομάδα, δεν είναι ομάδα ακτιβιστών. Όταν το λένε έχουν επιστημονική τεχνική, Αλλά υπάρχουν ε, βέβαια από πλευρά τεχνική επιστημονική κάποια θέματα στα οποία πάσχει αυτή η πρόταση. Όμως θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ αυτές διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ. Ε, εμείς ήμασταν αφανδόν αυτού του ρόλου μέσω κομισιών, μέσω, ε, όλων των υπηρεσιών Και Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα έγγραφο εργασία για να βοηθήσουμε τα κρατή-μέλη πριν την επόμενη συνάντηση στο ΟΗΕ. Να καταλάβει ο κόσμο, τι εννοεί με την πρότασή του ο ΠΟΗ. Όμω, θα πρέπει να δούμε για τα νέα κράτη-μέλη και το... Δεν θα είναι τόσο καλό να υπάρξει απόρριψη. Καλά. Μπορεί να γίνουν κάποιες ελάσσονες τροποποίησεις. Να, για παράδειγμα, κάπου αναφέρεται μέσα σε εκείνα τα έγγραφα ότι δεν υπάρχει υπερβολική δόση καναβιδόλης. Ναι, αλλά αν μιλούμε για ενεργή ουσία και αν σε μερικές περιπτώσεις έχει θεραπευτική χρήση εξορισμού από πλευράς χημίας, μπορεί να υπάρξει, μπορεί να νοηθεί υπερβολική δόση. Να, ένα θέμα το οποίο αν θέλουμε να περάσει το κείμενο πρέπει αυτό να διορθωθεί, αλλιώς δεν θα περάσει. Οπότε, προσταθήκατε να προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Μακάρι να ευδοκιμήσει η πρόταση. Θα είναι καλό για όλη την Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη στον ΟΗΕ να αγκαλιάσουν πρόταση, αλλά αυτό ακόμα δεν ισχύει. Τώρα, Γκαρό και κύριε η σχέση εγκληματικότητας και ναρκωτικών. Δηλαδή η διάθεση των ε, ναρκωτικών και της εγκληματικότητας ε, και κατά πόσο μπορούμε να πάμε σε πιο αποτελεσματικέ πολιτικές. Πρώτα-πρώτα δυστυχώς δεν υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ ε, αποτελεσμάτων και πολιτικής. Μα Βέβαια, ε, σε αυτό ε, είμαστε μοναδικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι περισσότερες εθνικές στρατηγικές αξιολογούνται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας. Και εμείς και εσείς. Ε, οι πρίσοι κρατών μελών μας βοηθούν να συστηματοποιήσουμε, να προτυπωποιήσουμε τις πληροφορίες και είμαστε μοναδικοί στον κόσμο ότι ακόμα και οι αξιολογίες γίνονται από εξωτερικούς αξιολογητές. Και τώρα πάμε στην ερώτηση της κυρίας Μπρικμόν. Εμείς αναλύουμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη των νομοθεσιών. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις γιατί είναι διαφορετικές οι ανομεστάξεις, αλλά σε τακτά διαστήματα κάνουμε αυτή την αξιολόγηση και ενημερώνουμε όλα τα κατημέλια. Γίνεται μελέτη όλων τι νομοθεσία έχουν, τι κριτηρία υπάρχουν. Όταν έχουμε αρνητικές συνέπειες βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά βοηθούμε τα κρατημέλη με ανάλυση, με πληροφορίες και έτσι τα κρατημέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία. Ας πούμε, παράδειγμα, για τις νέες ψυχότροπες ουσίες και επίσης κάτι άλλο, το θέμα της αποποινικοποίησης. Θα χρειαζόμουν ακόμα 15 λεπτά και ο πρόεδρος δεν θα με αφήσει κάποια άλλη φορά. Πάντως, άλλο νομιμοποίηση και άλλο αποποινικοποίηση. Και η πρώτη χώρα που εδώ και 20 χρόνια η θέση τα προσέγγιση ήταν η Πορτογαλία. Απέδωσε αποτελέσματα και αποδίδει ακόμα. Μετά από 20 χρόνια άσκηση της πολιτικής, αλλά πριν κλείσω, έχω να σας πω ότι αυτό που χαρακτηρίζει την πρωτοτυπία και τα αποτελέσματα της πορτογαλικής πολιτικής δεν είναι μόνο η αποποινικοποίηση, θεωρήθηκε η χρήση ναρκωτικών σαν κάτι που έχει συνέπειες για τη δημοσία υγεία, για τον κόσμο και είπαν ότι αντί να στέλνουν τον κόσμο στη φυλακή για μια απλή χρήση θα ήταν καλύτερα να τους ε, πάνε ε, προς κάποια προγράμματα θεραπείας και είναι πολύ μεγάλη αυτή η επένδυση και προς την ε, καταπολέμηση της ε, εμπορίας ναρκωτικών. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοστέλ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Πραγματικά κάθε λεπτομέρεια που μας δώσατε για τις δραστηριότητε σας ε, στον οργανισμό μας εμπλουτίζει. Σας ευχαριστούμε για τα πρωτογαλλικά σας, για τα ελληνικά σας. Βεβαίω για τα πρωτοκολλικά δεν, δεν μα ε, εκπλήξατε και τόσο πολύ, αφού η έδρα του οργανισμού σα είναι στην ε, Λισαβόνα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε και που μα βοηθήσατε με το χρόνο. Σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο και καλωσορίζουμε αμέσως τον διευθυντή του ΣΥΠΟΛ. Sí. Again, willkommen, Herr Schröder. Σας ε, καλωσορίζω. Έχουμε λοιπόν μαζί μας ε, τον Οργανισμό για την ε, Κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου. Να μην χάσουμε χρόνο, να του δώσουμε το λόγο τον κύριο Δέτλεφ Σρόιντερ, τον εκτελεστικό διευθυντή και όσοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, σας το λέω από τώρα, σας παρακαλώ, τηρήστε τα στενά χρονικά όρια που έχουμε και δυστυχώς ε, ζητούμε συγγνώμη και από τον κύριο Σρόντερ για το γεγονός ότι τον ε, καθυστερήσαμε, ότι βγήκαμε εκτός προγραμματισμού χρονικού. Θέλουμε να ακούσουμε την, ε, τα όσα έχει να μας πει για τον οργανισμό. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. many the members of the Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σα. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, ξέρω ότι έχετε και πίσω σα μια πολύ δύσκολη και κοπιαστική ημέρα. Πολύ σύντομα θα σα το πω. Θέλω σε κάποια σημεία μόνο να σταθώ κάπω πιο αναλυτικά. Θέλω ε, σήμερα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να φωτίσω, αν θέλετε, την ε, ανάγκη και τη σημασία που έχει η κατάρτιση στον τομέα του, της επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Τι είναι το ΣΥΠΟΛ. Είναι η Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της ε, επιβολής του νόμου. Παλαιότερα ήμασταν ε, υπεύθυνοι μόνο για τις αστυνομικές αρχές. Πλέον όμως εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε και εισαγγελείς, συνοριοφύλακες. Στην Ουγγαρία είναι η έδρα μας. Συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη. Σε 26 έχουμε εθνικές, σε 26 κράτη-μέλη έχουμε ε, εθνικές μονάδες και ε, συνεργαζόμαστε και σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Συνεργαζόμαστε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα με τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η εντολή μας, τι κάνουμε με βάση την εντολή μας. Υποστηρίζουμε ε, τις ε, εγχώριες δραστηριότητες, προγράμματα ανταλλαγής, Προωθούμε την αμοιβή αναγνώριση στον τομέα της, της κατάρτισης, στον τομέα της επιβολής του νόμου. Αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε αναλυτικά προγράμματα και ε, καθορίζουμε και χαρτογραφούμε ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης των κρατών μελών. Δρούμε συμπληρωματικά προς τα όσα ήδη γίνονται δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Τι έχουμε πετύχει το 2018. Το 2018 εκπαιδεύσαμε πάνω από 29.000 αξιωματικούς συμμετούχους από την Ευρώπη και από τρίτες χώρες. Και το ποσοστό ικανοποίησης είναι υψηλό. 94% των συμμετεχόντων στους κύκλους εκπαίδευσής μας, κατάρτισής μας, ε, δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι. Εμείς υποστηρίζουμε όλες τις βασικές ενωσιακές προτεραιότητες, δηλαδή σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, αντιτρομοκρατία, παράτυπη μετανάστευση και κυβερνοέγκλημα για το οποίο θα σας πω αργότερα περισσότερα στοιχεία. Εδώ βλέπετε πώς ε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια η συμμετοχή στη ΣΥΠΟΛ. Ξεκινήσαμε το 2009 με 2.000 περίπου συμμετέχοντες στις δραστηριότητες μας. Πέρσι πάνω από 29.000 συμμετέχοντες είχαμε. Και για φέτος ε, εκτιμούμε ότι θα καταρτήσουμε πάνω από 35.000 συμμετέχοντες από τα κράτη-μέλη. Αυτό που εσάς σας ενδιαφέρει είναι ε, ότι έχουν όλα αυτά γίνει με περίπου ε, σταθερό προσωπικό και σταθερό προϋπολογισμό. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου ουσιοδός δηλαδή ο προϋπολογισμός μας ή το προσωπικό μας. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση από τα κράτη-μέλη, από όλα τα κράτη-μέλη, και νομίζω ότι πλέον δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον ε, στη ζήτηση από τα κράτη-μέλη αν οι δραστηριότητες ε, ε, μάλλον οι δραστηριότητε μα, τα αιτήματα που, ζητούμε, που δεχόμαστε από τα κράτη-μέλη έχουν τριπλασιαστεί. Δεν ξέρουμε πώ θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση. Τι κάνουμε λοιπόν. Έχουμε πάνω από 100 ε, εσωτερικές ε, όπου συμμετέχουν ε, συμμετέχουν αξιωματούχοι από τις αρχές των κρατών μελών. Ε, έχουμε online course, τα webinars δηλαδή, ε, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο. Ζωντανά μέσω διαδικτύου εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε πάνω από χίλιους συμμετέχοντες. Μπορούμε κάθε φορά να εξυπηρετούμε. Έχουμε και τις ανταλλαγές SIPOL που, που δίνουν τη δυνατότητα σε έναν αξιωματούχο να, να πάει σε μια άλλη χώρα για να λάβει πραγματική εμπειρία για το ποιε είναι οι συνθήκε που επικρατούν σε μια άλλη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ενισχυθεί η συνεργασία. Αν δηλαδή πάει κάποιο άνθρωπο σε μια άλλη χώρα ε, ή καλείται να συνεργαστεί με συναδέλφους του από άλλη χώρα, τότε πραγματικά είναι μεγάλη αξία του να ξέρει ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην αρχή στην άλλη χώρα. Πέραν αυτών, των ε, κύκλων κατάρτισης για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κύκλους και για τρίτες χώρες. Πέρσι συνεχίσαμε ένα ε, project αντιτρομοκρατίας με χώρες από τη Μέση Ανατολία και τη Βόρη, Βόρεια Αφρική. Τις βλέπετε εδώ τις χώρες στα αριστερά. Είναι ένα εργαλείο για, που ενισχύει και τον αντιτρομοκρατικό διάλογο με αυτές τις χώρες και ε, καταβάλουμε ε, πολλές ε, προσπάθειες και ε, με τις χώρες αυτές, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο ε, που ενισχύει τη συνεργασία των αντιδρομοκρατικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ένα άλλο project που τρέχουμε είναι με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, για με τις οποίες υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίες, τις οποίες υποστηρίζουμε και ε, επιχειρησιακά και οικονομικά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το project είναι ε, οι έξι χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δυτικών Βαλκανίων να έρθουν σε επαφή με τα κράτη-μέλη όταν ακριβώς χρειάζονται ε, βοήθεια και αυτό μπορεί πάντοτε να γίνεται με πολύ καλό συντονισμό. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, πρέπει να σας πω αυτά που σας είπα ε, εμπίπτουν μέσα στην ε, αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, ανάγκες στρατηγικής κατάρτισης. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά αυτό που είναι καινούριο είναι ότι κάναμε μια ανάλυση του ποιοι είναι οι τομείς, ποια είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν, πού υπάρχει ζήτηση, πού πρέπει να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τον δικό μου οργανισμό, αλλά και άλλου οργανισμούς. Ποια είναι ακριβώς, ποιες είναι οι θεματικέ ενότητες στις οποίε πρέπει να ε, επικεντρωθούμε. Και από τις συνεντεύξεις που κάναμε με πάνω από 500 εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη, βλέπετε εδώ ποιοι είναι οι τομείς ε, στου οποίου πρέπει να ε, επικεντρωθούμε. Του ρωτήσαμε Πού θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά, πού υπάρχουν χάσματα, πού υπάρχουν παραθυράκια, πού πρέπει εμείς να παρέμβουμε για να σας βοηθήσουμε. Μιλάμε για μυστικές προφορίες, κυβερνοασφάλεια, κυβερνοέγκλημα. Αυτή είναι ε, η βασικότερη τομή στους οποίους θα επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να σας τονίσω ότι ό,τι κάνουμε εμείς επιχειρησιακά το κάνουμε πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους ε, οργανισμούς εταίρους μας. Και εδώ βλέπετε μόνο κάποιους από αυτούς μπορώ να σας πω επίσης ότι ε, συνεργαζόμαστε και με την EMCDDA, αλλά με την Europol για παράδειγμα, το, για το 75% των ε, δραστηριοτήτων μας κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Europol, Eurojust, Eurolisa, ε, εργαλεία διαδικτυακά. Όλα αυτά μας βοηθούν γιατί εμπλουτίζουμε και με τα δικαστικά, για παράδειγμα, ζητήματα, αλλά και με τη Frontex. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία επιχειρησιακή και λειτουργική. Επίσης, κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, είναι κάποια βασικά στοιχεία. Από στρατηγική άποψη, αποφασίσαμε να κάνουμε και μια διασφάλιση ποιότητας. Έχουμε πλέον, ε, τηρούμε πλέον ε, το πιστοποιητικό ISO 9001, γιατί ε, πλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις ε, ε, απαιτήσεις που έχει πλέον ο, και τα πρότυπα του κλάδου και ε, πραγματικά είναι ε, ύψης της ποιότητας η κατάρτιση που παρέχουμε. Και όπως είπε και ο συνάδελφος από το e MCDDA, μπορώ να σας πω και εγώ ότι η εκτέλεση του προπολογισμού μας ανήλθε σε επίπεδα άνω του 95%, η εκτέλεση το 2018 όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας ανήλθε σχεδόν στο 98% και αυτό είναι ένα πολύ ε, θετικό σημάδι γιατί δείχνει δημοσιονομική πειθαρχία από τον πλευρά μας. Μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε ο μεγαλύτερος ε, οργανισμός, έχουμε 32 μόνιμα μέλη προσωπικού, αλλά έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και πρέπει να τους ευχαριστήσω γιατί χωρίς την προσήλωση όλων των μελών της ομάδας μας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε επιτύχει τόσο καλά αποτελέσματα. Τώρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε ήδη από τώρα και για το, 2000, ε, για το, για το 2019 δηλαδή. Για το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2019, για ε, μια καθοδήγηση αν θέλετε, ποια είναι η πόρη που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε ζητήσει για το 2019 12 εκατομμύρια προϋπολογισμό και εδώ ε, βλέπετε ότι δεν είναι και ο μεγαλύτερος οργανισμός ο δικός μου. Έχουμε ζητήσει 40 προσωρινούς συμβασιούχους. Ε, λάβαμε τελικά ε, με βάση τα αιτήματά μας 9,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας εδώ και 10 χρόνια κάθε χρόνο. Και έχουμε 32 συμβασιούχους και ε, εργολαβικούς. Και Έχουμε λάβει και για τα δύο project που σας ανέφερα νωρίτερα 8,9 ε, εκατομμύρια ευρώ για την τριετή διάρκεια όμως των προγραμμάτων αυτών. Ποια θέματα ε, μας απασχόλησαν φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Αντιτρομοκρατία και όλα τα συναφή όπως αναφέρατε και εσείς ε, στη συζήτηση για τη Eurojust. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα καυτό για τα κράτη-μέλη. Από, από την δική μας σκοπιά και με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από την Europol υπάρχουν δύο βασικές ε, τάσεις, η Ισλαμική τρομοκρατία και η ακροδεξιά τρομοκρατία. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται πάρα πολύ με τους ε, εγχώριους ε, τρομοκράτες, δηλαδή ανθρώπους που έχουν ε, ζήσει, γεννηθεί ε, σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, όμως τελικά ριζοσπαστικοποιούνται και γίνονται τρομοκράτες και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, ξένοι μαχητές ε, που επιστρέφουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Εκεί επίσης έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε. Θέλουμε να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι της κοινότητας για να, για να μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο για το τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους επιστρέφοντες. Γιατί ε, πολλές φορές ε, μπορεί να γνωρίζουμε αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κάποιον που έχει επιστρέψει. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια ανταλλαγή ε, πρακτικών αν θέλετε. Επίσης μας απασχολεί η ριζοσπαστικοποίηση, η απο-ριζοσπαστικοποίηση, ποια είναι η σημασία και η συμβολή των social media σε όλα αυτά. Πρέπει εμείς να μάθουμε περισσότερα για τις διασυνδέσεις ανάμεσα στην τρομοκρατία και το έγκλημα. I Επίσης, να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος από την ε, Eurojust. Ποια, ποιες είναι οι βασικές, βασικές προκλήσεις. Κυβερνοέγκλημα ε, είναι πράγματι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Δύο στοιχεία θα σας δώσω. Η, η Κομισιόν θεωρεί ότι ήδη 50% όλων των αδικημάτων που διαπράττονται είναι κυβερνοεγκλήματα. 50% των εγκλημάτων που διαπράττονται σε, ε, στα κράτη-μέλη. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ότι έως το 2020 θα έχουμε απόλυες 3 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέονται ε, οικονομικών ζημιών, δηλαδή που, με, που θα συνδέονται με, την, με το κυβερνοέγκλημα. Αυτά τα, ε, μπορείτε να σας ζητήσετε σε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και με την Europol. Εδώ λοιπόν η κοινότητε και οι αρχές επιβολή του νόμου πρέπει να κάνουν άλματα για να βελτιώσουν την κατανόησή τους και τις ψηφιακές τους δεξιότητε. Και ερώτημα, είμαστε έτοιμοι. Να σας θέσω μόνο κάποια θέματα. Δίκτυα 5G που θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Το διαδίκτυο των πραγμάτων. Ο όγκος των δεδομένων που θα πρέπει να τίθενται σε επεξεργασία θα εκραγεί, θα εκτοξευτεί και ήδη τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν πώς μπορούν τόσα πολλά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή να τα επεξεργάζονται. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Αυτοκίνητα χωρί οδηγού. Συζητιέται συχνά. Κάποια στιγμή θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό έχει σημασία και για τι αρχέ επιβολή του νόμου γνωρίζουμε, έχουμε τις ε, επαρκείς γνώσεις, πώς ακριβώς θα λειτουργούν αυτά τα αυτοκίνητα με τους υπολογιστές. Τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται πολλή συζήτηση, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που αφορά τις, άρχες, τις αρχές επιβολές του νόμου, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικές γνώσεις στους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Πώς ακριβώς θα την αξιοποιήσουν αν δεν την γνωρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ αυτό που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Κρυπτονομίσματα, όταν μιλάμε για οικονομικές έρευνες. Είναι ήδη πρόκληση όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κρύψουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά την ε, πορεία των χρημάτων και των κρυπτονομισμάτων. Και αυτό επίσης απαιτεί συγκεκριμένε δεξιότητες. Ψευδείς ειδήσει, χειραγώγηση. Για εσάς που είστε και πολιτικοί δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και εκεί νομίζω ότι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν είναι πάντοτε επαρκώ προετοιμασμένε. Και νέα πληροφορικά συστήματα μηχανοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαλειτουργικότητα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί πρέπει να ε, όλοι αυτοί που θα τα χειρίζονται αυτά τα νέα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να, έχουν τις ε, επαρκείς δεξιότητες και γνώσεις, να ξέρουν τι μπορούν, σε, σε τι μπορούν να τα, να τα αξιοποιήσουν αυτά τα νέα εργαλεία και σε τι όχι. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ε, επαρκής και κατάλληλη κατάρτιση. Ψευδείς ειδήσει, κίνδυνοι για εκλογέ. 61% των Ευρωπαίων ήδη ανησυχούν για τη χειραγώγηση μέσω κυβερνοεπιθέσεων. 59% ανησυχούν σχετικά με ξένους πράκτορες και εγκληματικέ ομάδες που επηρεάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Και όχι μόνο στο Facebook και άλλες πλατφόρμες με ποσταρίσματα ψευδών ειδήσεων. Άμα δείτε τις ε, τρέχουσες συζητήσεις για τις, για τις ειδήσει deepfake όπου έχουμε να κάνουμε ε, με δηλώσεις που δεν μπορεί κανείς να διακρίνει αν είναι αληθινές ή όχι, μέσω χειραγωγημένων, παραποιημένων βίντεο για παράδειγμα. Και εδώ πρέπει οι αρχές επιβουλές να έχουν τις ικανότητες να τις αντιμετωπίζουν αυτές τις υποθέσεις. Εμείς λοιπόν στη ΣΥΠΟΛ τι κάνουμε, έχουμε κάνει τη Cyber Academy και εκεί εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε αξιωματούχους των κρατών μελών. Έχουμε μοντέρνα τεχνολογία με την οποία μπορούμε να εκπαιδεύουμε τους αξιωματούχους αυτού. Και βλέπω κάποιες φορές ε, κάποια κράτη-μέλη να μην έχουν ένα αντίστοιχο κέντρο για την ε, αντιμετώπιση του κυβέρνου εγκλήματο. Όποιος λοιπόν έχει τέτοιες, ε, τέτοια επιθυμία, εμεί έχουμε συλλέξει πολλέ γνώσει και πολλή εμπειρία Όταν ρωτήσαμε από τα κράτη-μέλη πόσου πιστεύετε ότι χρειάζεται να καταρτιστούν στον τομέα του κυβέρνου εγκλήματο, η απάντηση η συνολική ήταν 140.000. Ωστόσο, το κυβέρνο έγκλημα είναι μία πλευρά μόνο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε και τι παραδοσιακέ. Ναρκωτικά, νέε ψυχοδραστικές ουσίε, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και αντίστοιχα εγκληματικά δίκτυα, διακίνηση ανθρώπων και όλα τα άλλα ζητήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουν οι αρχέ επιβολή του νόμου. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται δεξιότητε, προσόντα πραγματικά στι ε, αρχέ τη επιβολή του νόμου. Γιατί οι πολίτε πραγματικά αξίζουν να έχουν τέτοιε ε, δεξιότητες, τέτοιες αρχές ε, του νόμου, γιατί στα χέρια τα δικά τους είναι τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα των ε, πολιτών. για να γίνει αυτό χρειάζεται οι αξιωματούχοι να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Ποιος είναι ο ρόλος της ΥΠΟΛ λοιπόν. Εμείς θέτουμε σε πράξη, στην πράξη τα νομικά εργαλεία και τις πολιτικές. Τι κάνουμε δηλαδή, δίνουμε στον κόσμο, στου, το, ανθρώπους που εργάζονται στις αρχές επιβουλής του νόμου, πώς μπορούν, ποια, τους δίνουμε να καταλάβουν ποια είναι τα εργαλεία, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, πού μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και δεν μιλάμε μόνο για τις κοινέ ε, ε, ομάδες ερεύνης. Έχουμε μια σειρά από εργαλεία, εδώ και 20 χρόνια έχουμε ε, συλλέξει εμπειρία. Ε, πολλές φορές, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι οι εισαγγελικέ και αστυνομικέ αρχέ κάνουν την ίδια ακριβώ δουλειά, κάνουν τις ίδιες έρευνες χωρίς να το γνωρίζουν πολλές φορές. Επίσης, συμβάλλουμε ε, και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων, ε, του ανθρωπίνου δυναμικού. Συμμετέχουμε και συμβάλλουμε και στην δημιουργία μιας κοινή ευρωπαϊκής κουλτούρας για την επιβολή του νόμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η εμπιστοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών των κρατών μελών είναι ουσιαστική σημασίας για την καλή συνεργασία. Και τέλος αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και ο οργανισμός μας να έχει τον επαρκή προϋπολογισμό και επαρκείς πόρους. Γιατί όπως είπα δεν έχουμε ε, καμία αύξηση τα τελευταία χρόνια ε, στον προϋπολογισμό μας και στο προσωπικό μας τα καταφέραμε, αλλά δεδομένου τη ζήτηση που θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, ελπίζουμε να έχουμε και τη δική σας στήριξη, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό μας για να μπορέσουμε με τη σειρά μας να παρέχουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ και τώρα η σειρά των βουλευτών να κάνω κάποιε ερωτήσει ε, Αν θέλετε να μα ζητήσετε το λόγο. Θα είστε οι η κυρία Τρουγκάριου είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα πάρα πολύ συνοπτική. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω. Δεν ε, ξέρω αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά μπορείτε να απαντήσετε και γραπτά και να μιλήσω ρουμάνικα τη γλώσσα μου. Πρόσφατα στη Ρουμανία είχαμε διάφορες περιπτώσεις και κυρίως η υπόθεση Καρακάλ, την οποία κάλυψε και ο Διεθνής Τύπος για απαγωγές και δολοφονίες εφήβων. Τέτοιες υποθέσεις σχετίζονται με διακίνηση ατόμων και σχετίζονται με το γεγονός ότι η ρουμανική αστυνομία χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, κατάρτιση, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι στη διακίνηση ανθρώπινων ε, ανθρώπων 67% είναι γυναίκες και κορίτσια και στην κορυφή των, της λίστας ε, είναι πέντε χώρες από τις χώρες των Βαλκανίων ε, και της Κεντρικής Ευρώπης, ε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν προβλήματα σε αυτές τις χώρες. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να κάνω είναι το εξή. καταρχά. θα ήθελα να μου πείτε τον αριθμό των καταρτήσεων σε ό,τι αφορά την διακίνηση ανθρώπων τι οποίες έχει συμμετέχει η Ρουμανία τα τελευταία χρόνια. Έγιναν τέτοιες ε, καταρτήσεις για τη Ρουμανία ιδιαίτερα και ειδικά ή για άλλες χώρες τις οποίες και να συμμετείχε η Ρουμανία. Το δεύτερο το κέντρο σας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων. Να βοηθήσει, για παράδειγμα, την αστυνομία της Ρουμανίας για να εκπαιδευτεί σωστά για την καταπολέμηση τέτοιων δικτύων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα για το λόγο εσείς κυρία Καλλιλάντ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και για την ε, παρουσίασή σας, την παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τα θέματα για το κυβέρνο έγκλημα. Πάνω από το ίμιση των ε, εγκλημάτων σήμερα, όπως είπατε, έχουν να κάνουν το κυβέρνο έγκλημα. Αναφερθήκατε σε διάφορα είδη εγκλήματο. Εγώ θέλω να σα ε, ρωτήσω για την ε, βία στο διαδίκτυο. Είναι κάτι το καινούριο, καινούριο, καινούρια μορφή βίας. Στόκινγκ, παρενόχληση, ό,τι και να σημαίνει. Είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί τα θύματα συνήθω είναι ιδιαίτερω ευάλωτα και διστάζουν να καταγγείλουν τα εγκλήματα στι αστυνομικέ αρχές και σύμφωνα με την εμπειρία μας ε, οι αστυνομικοί δεν τα παίρνουν και πάντα στα σοβαρά. Δυστυχώς όμως η βία online στο διαδίκτυο σήμερα φαίνεται ότι είναι λιγότερο σημαντική θεωρείται σε σχέση με την ε, κοινή μορφή και οι πιο συνήθεις, ε, τα πιο συνήθι θύματα είναι οι γυναίκες, ε, παιδιά και οι μετανάστες. Έχετε λοιπόν συμπεριλάβει αυτή τη βία στο διαδίκτυο στα προγράμματα εκπαίδευσης και διακρίνεται κάποιο ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Κάποια άλλη ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Αν όχι. Κύριε Σρόντερ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Και καταρχάς το πρώτο ζήτημα για το THP και για τα ε, θύματα, παιδιά και γυναίκες ε, και σε ό,τι αφορά την ε, παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης στη Ρουμανία, στη Ρουμανική αστυνομία. Μπορώ να σας δώσω πληροφορίες, αλλά να σας πω τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά επικεντρωνόμαστε στο θέμα αυτό. Το για την προστασία των θυμάτων και θα σας δώσουμε λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία για τις ρουμανικές αρχές. Να σας πω ότι συχνά οι ρουμανικές αρχές μας προσέγγισαν και ε, μας ζητούσαν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάποιες συγκεκριμένε υποθέσεις σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ε, ανθρώπων. Το δεύτερο θέμα για την βία στο διαδίκτυο. Είμαι ενήμερος για το θέμα αυτό και αντιλαμβάνομαι ότι σε ορισμένε περιπτώσει τα θύματα ακόμα και έχουν αυτοκτονήσει λόγω τη βία αυτή. Ω τώρα το έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μα έμεσα, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε οι ερευνητέ να χρησιμοποιήσουν καταρχά την τεχνολογία, γιατί σε πολλέ περιπτώσει δεν μπορούν καν να εξετάσουν τα τεκμήρια, δεν κατέχουν την τεχνολογία και γι' αυτό είναι κάπω διστακτική. Αλλά θα χαρώ να το κοιτάξω πιο ενδελεχώς το θέμα αυτό. Να δούμε δηλαδή και τα κράτη-μέλη θα μας ζητήσουν συγκεκριμένα σε εκπαίδευση. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει ζητήσει κάποιο κράτος μέλος συγκεκριμένα να υπάρξει εκπαίδευση στο θέμα αυτό. Γιατί συχνά ξέρετε οι ερευνητέ δεν είναι σε θέση, δεν έχουν τα προσφότα για να καταγράψουν τέτοια περιστατικά. Και ως τώρα εκεί εργαζόμαστε, σε αυτό το τομέα, στην καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των ερευνητών, αλλά με χαρά να το συμπεριλάβω στο θέμα αυτό και στις μελλοντικές μας προτεραιότητες. Ήταν μεγάλη η σημερινή ημέρα και έχουμε και ακόμα ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η παρουσία του κυρίου Σρόντερ ήταν πολύ επόφελη. Τον ευχαριστούμε για την παρουσίασή του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια. And if you spare some additional... Και τώρα, αν έχετε ακόμα λίγο κουράγιο, ό,τι σας έχει απομείνει... Skills to the lengthy and wait. Μετά από την ε, μεγάλη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής μας, να κοιτάξουμε το επόμενο θέμα. which is the presence here of uh, candidate. Yes. Yes. Yes, yes. Πρόκειται για την εφαρμοστική απόφαση έγκρισης της σύναψη της συμφωνίας μεταξύ Eurojust και Σερβία. Έχω αναλάβει ο υπεφαινόμενο να είμαι ο και έχει προηγηθεί διαδικασία διαβούλευσης για αυτήν την συμφωνία. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν συναυθεί στο παρελθόν από την Eurojust με την Αλβανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, Ενωμένε Πολιτείες, Ελβετία, Μολδαβία και άλλες χώρες. Είναι πολύ κοντινή η καταληκτική ημερομηνία και συμφώνησαν οι συντονιστές τον Ιούλιο ότι θα πρέπει να έχουμε προσταθμένη διαδικασία όσον αφορά την έγκριση. Επομένως δεν θα έχουμε διαδικαστικές ε, τροπολογίες. Οπότε αποφασίστηκε ότι ο πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ θα αναλάβει την εισήγηση. Και η προθεσμία για την διαβούλευση ε, που κρατά τρεις ε, μήνες θα εκπνεύσει στις 10 Οκτωβρίου. Τώρα δηλαδή, την επαύριο. Οπότε θα δώσουμε τώρα ε, ξανά στο εκπρόσωπο του γύρω λόγο για να μας παρουσιάσει αν θέλει κάποιες ε, διευκρινήσεις, κάποια σημεία. Έχουμε τον Αντιπρόεδρο κ. Μάιερ Κάβλε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ αγαπητοί κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω άλλη μια συμφωνία δικαστικής συνεργασίας που συνήφθη από την υπηρεσία μας. Και αυτές οι συμφωνίες μας ε, δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί για την ε, αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Όπως είπε ο Πρόεδρός μας, ε, υπάρχει ωφέλεια από αυτές τις ε, συμφωνίες, είναι εκθετική η ωφέλεια. Και έχουμε επίσης και τους εισαγγελίες που είναι πέσπασμένοι από αυτές τις χώρες στην Χάγη. Και θέλουμε στα Δυτικά Βαλκάνια να εφαρμοστεί η στρατηγική μας, να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και ασφαλεία επίσης. Θέλουμε να θωρακιστεί το κράτος δικαίου, να βοηθήσουμε στα Δυτικά Βαλκάνια τις ε, μεταρρυθμίσεις. Στα πλαίσια των προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αλλά βέβαια και έτσι καταπολεμούμε το έγκλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνεργαζόμενες χώρες. Ε, προστασία δεδομένων και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από εμά και από τους ε, εταίρους μας. Το ίδιο ισχύει και για τη Σερβία και πρώτα-πρώτα όλα τα αιτήματα της ε, Eurojust για προστασία δεδομένων, τα, όλα αυτά τα δέχτηκαν οι Σέρβοι και τροποποίησαν τον ε, σχετικό τους νόμο επί τη βάση αυτής της συμφωνίας και ήδη έχει αρχίσει η φάση της εφαρμογής και έδειξαν ε, ανοιχτό πνεύμα για όλες μας τις προτάσεις. Άρα, έχουμε τώρα ένα στεγανό σύστημα προστασίας δεδομένων και όπως προαναφέρθηκε θα γίνεται ετήσια αναθεώρηση ούτως ώστε να μην χαμηλώσει ο πύχης. Τώρα, ο προστάμενος της ε, εισαγγελίας στην ε, Σερβία απέδειξε ότι είναι συνομιλητής ε, αξιόπιστος και ήδη έχουν γίνει κοινέ ε, έρευνες. Το 2018 η Σερβία ήταν στη δεύτερη κατάξη όσον αφορά τις χώρες που συνεργάζονται μαζί μας για τις υποθέσεις, τον αριθμό των υποθέσεων. Και μόλις αποσπαστεί η εισαγγελία στην υπηρεσία μας θα έχουν περισσότερη συνεργασία. Ήδη, ήδη ο προς τα έχει αρχίσει τις σχετικές ενέργειες. Και αν εγκρίνεται αυτή τη συμφωνία, τότε θα το συνδυάσουμε και με την αστυνομική συνεργασία. Με αυτή τη δικαστική συνεργασία. Οπότε έτσι θα θρέξει το κράτος δικαίου και θα πλαισιώσουμε τις προσπάθειες που γίνονται για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και με αυτή τη συμφωνία δεν θα έχουμε ενέργειες σχετικές με τη Σερβία από οποιοδήποτε κράτος μέλος μεμονωμένα, αλλά από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό. Και η Σερβική Αγγελία και το Υπουργείο Ιστορικών είπαν ότι ό,τι προβλέπει η συμφωνία θα τα τηρήσουν, τα εφαρμόσουν και αυτό θα ωφελήσει και τους Σέρβους αλλά και τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτούς όλους τους λόγους σας τον Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για όσα μας είπατε. Όλα αυτά. Ε, γίνονται αυτή η διαδρομή τέλο πάντων εξελίχθηκε σε μεταβατική φάση εν των ευρωεκλογών. Πάντως, εμείς θα πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό της διαδικασίας έγκρισης. Να ολοκληρωθεί ταχαίως η διαβούλευση. Να μην έχουμε ε, τροπολογίες, διαδικαστικές, να έχουμε την λεγόμενη απλουστευμένη διαδικασία. Έχετε κάποια ένσταση, κάποια παρατήρηση σε σχέση με αυτά που προτείνουμε ως διαδικασία. Όχι, από ό,τι φαίνεται, οπότε εγκρίνεται ως έχει... Επομένως, απλώς το ισχύ, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου θα σας παρουσιάσω το σχέδιο κειμένο ο υποφαινόμενος ως πρόεδρος και εισηγητής 24 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και τον Οκτώβριο η δυνατόν θα γίνει η έγκριση στην Ολομέλεια οπότε έτσι θα έχουμε τηρήσει αυτό το αυστηρό χρονοδιόγραμμα. Αν δεν υπάρχει ένσταση, σας ευχαριστώ. Hey, tomorrow, do for the afternoon session. Tomorrow, Αύριο θα γίνει ψηφορία αύριο το πρωί. Για σε ελάτε έγκυρα. Και πέστε το ότι χρειάζεται η κάρτα και η ηλεκτρονική ψηφορία. Ευθύσαμε στην αρχή της πρωινής συνεδρίας. Τα λέμε αύριο.